Right. Uh, um, uh, Καλώς ήρθατε. Κάνω μια εισαγωγή για το θα κάνουμε. 27 Οκτωβρίου ο πρόεδρος Μπαρόσο ανακοίνωσε κάποιες αλλαγές στα φυλάκια. δύο επιτρόπων που εμπίπτουν στην εντολή της Επιτροπής μας. Ρεν και Σέμετα, δηλαδή των δύο επιτρόπων αυτών. Ο Επίτροπος Ρεν έχει ε, αποκτήσει και άλλες εξουσίες, έγινε και αντιπρόεδρος και έχει και άλλους ρόλους και άλλη δουλειά και άλλα μέσα στη θέση του για να βοηθήσει τον πρόεδρο με το έργο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ε, οικονομική διακυβέρνηση, συνόδους κορυφής, ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης. Τα υπόλοιπα λέω μετά. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα βάσει του άρθρου 166 του εσωτερικού κανονισμού. Μαζί με το παράρτημα 27.2 σι λατινικό, καλούμε τον Επίτροπο να εμφανιστεί προ της αρμοδίας επιτροπής πριν να αναλάβει τα καθήκοντά του, καθήκοντά τους. Αυτό κάνουμε λοιπόν, καλέσαμε τον Επίτροπο, θα διεξαχθεί η ε, ακρόαση. Α, άλλη διαδικασία προβλέπεται έγιναν ανακοινώσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Θα δώσουμε λοιπόν στον Όλη ένα 20 λεπτό. Θα μας κάνει μια παρουσίαση η οποία φαντάζομαι ότι συμπεριλαμβάνει και κάποια ενδιαφέροντα έγγραφα. Μετά θα ακολουθήσουν όλα τα απαντήσει. Είναι πολύ περιορισμένο το χρονικό διάστημα, ένα λεπτό για ερώτηση, δύο λεπτά για απάντηση. Ίσως υπάρχει επικάλυψη, αλληλεπικάλυψη των ερωτήσεων. Άρα θα ακούσουμε από την αρχή σε ομάδες των τριών τις ερωτήσεις. Τρεις ερωτήσεις και μετά ένα εξάλεπτο για απάντηση στις ερωτήσεις. Και άρα νομίζουμε ότι τα χειριστούμε καλύτερα έτσι. Αντί να έχουμε ένα τόσο στενό πρόγραμμα ερωτήσεων-απαντήσεων, αν ξεπεράσει κάποιος το χρόνο του, ε, δεν θα μας περισσέψει χρόνο στο τέλος. Οι συνέπειες θα πληρωθούν από τους μεταγενέστερους ομιλητές και θα κρατάω και λογαριασμό ε, για τις τρεις ομάδες να μην μιλήσει περισσότερο μια ομάδα πολιτικής βάρος της άλλης. Τούτων λεχθέντων, Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Σάρουν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να συζητήσουμε σημαντικότατα θέματα μαζί σας σήμερα. Ο λόγος για την ανταλλαγή απόψεων, ο τυπικός, είναι να σας δώσω τη δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήσεις σχετικά με την αλλαγή του χαρτοφυλακίου μου. Αυτό που σα εξήγησε Σάρων. Με τα χαράς λοιπόν να το κάνω αυτό και να απαντήσω και συγκεκριμένε ερωτήσεις επί του θέματος. Ταυτόχρονα δράτω με τη ευκαιρία να αναφερθώ στο λόγο για τον οποίο έγινε αυτή η κίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς θα βγούμε από την οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση που μαστίζει την Ευρώπη. Θέλω να μιλήσω και για τη στρατηγική που επιδιώκουμε για να πετύχουμε το στόχο μας να επανέλθει η Ευρώπη σε βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Αυτή ήταν η ουσία της αποφάσεως της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής Έχω και κάποια ε, πράγματα να σα περιγράψω, παρουσιάσω και κάποιους πίνακες και γραφήματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου. Ο ρόλος μου τώρα, που έγινε αντιπρόεδρος για οικονομικά και νομισματικά θέματα και για το ευρώ. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Όταν μιλώ για τον αντιπρόεδρο στο τρίτο ενικό δεν είναι γιατί είμαι μεγαλομανής αλλά αναφέρομαι στον αντιπρόεδρο ως θεσμό. Και δεν μιλώ για μένα προσωπικά, μιλάμε για μια θεσμική μεταρρύθμιση βλέπετε. Όταν ο πρόεδρος Μπαρόσο σας ανακοίνωσε ότι θα με διορίσει αντιπρόεδρο, είπε ότι ε, εμπεριέχει πραγματική πτυχή, ρεαλιστική πτυχή, αύξηση εξουσιών, αλλά επίσης υπήρχε και συμβολική πτυχή. Θα εστιαστώ επί των αυξημένων ευθυνών που συνεπάγεται αυτή η θέση εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά διάφορους ε, τομείς πολιτικής. Μεταξύ άλλων τι καλύπτω. Επίσημες προειδοποίησεις προς τα κράτη-μέλη σύμφωνα με τα προληπτικά μέτρα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης συστάσεις προς το Συμβούλιο μπορούν να απευθύνονται για κυρώσεις δυνάμει της νομοθεσιας Sixpack και εδώ καλύπτουμε τις διευρυμένες δυνατότητες εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις χώρες της Ευρωζώνης. Στα πλαίσια των προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας προς την Ευρωζώνη ή προς τις χώρες εκείνες Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω οικονομικής αστάθειας και εκεί χρειάζεται δράση από την Ευρωζώνη. Αυτή η εξουσία που δίνεται συνεπάγεται το ότι σε αυτού του τομεί ο αντιπρόεδρο που είναι υπεύθυνο για οικονομικά νομισματικά θέματα και το ευρώ μπορεί στο μέλλον, δρώντα εν συνεργασία με τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υιοθετεί αποφάσει. Αποφάσει εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν σώμα. Αυτό δίνει σημαντικό βαθμό αυτονομία στον αντιπρόεδρο το επιτρέπει ή τι επιτρέπει να εξασφαλίζει ουδέτερη οικονομική ανάλυση υψηλής ποιότητας που θα διαμορφώνει τις πολιτικές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει σαφή διαχωρισμό λοιπόν τώρα μεταξύ οικονομικής αναλύσεως που στηρίζει τις αποφάσεις όπου εκεί ο Αντιπρόεδρος έχει πολύ σημαντικό βαθμό αυτονομίας. Απ' την άλλη, διαχωρίζεται από τις πολιτικές ε, αποφάσεις που παίρνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαν σώμα. Υπάρχει και μεταφορά ευθυνών όσον αφορά το Eurostat στον Επίτροπο Σεμέτα. Αυτό τι συνεπάγεται. Συνεπάγεται διαχωρισμό πάλι ευθυνών για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων και για ανάλυση από τη χρήση των στοιχείων για οικονομικούς υπολογισμούς και αναλύσεις που είναι δική μου ευθύνη. Δράτω με τη ευκαιρία να ευχαριστήσω τη Eurostat. Έξοχη συνεργασία. Πολύ ψηλή ποιότητα των εργασιών τη. Και θα μου λείψει αυτό το τμήμα του παλαιού μου χαρτοφυλακίου. Απ' την άλλη, αποφασίστηκαν αυτά σε συμφωνία με τα αιτήματα για την τυπική ανεξαρτησία της Eurostat. Ακόμα και αν στην πράξη δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα όσον αφορά την εξαρτησία της Eurostat. Πριν από δύο ώρες περίπου, υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πακέτο για την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση. Εδράζεται εντός της στρατηγικής προσεγγίσεως για την Ευρώπη για το 2020. Κάτι που εγκρίνατε αφού το συζητήσατε. Και ετοιμάζεται και σχετικά ψηφίσματα. Και διαμορφώνει τη γενική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Στην ακρόαση για την ανάλυση των καθηκόντων εδώ και δύο χρόνια είπα ότι δεσμεύομαι να δημιουργήσω οικονομία της αγοράς που θα είναι κοινωνική και ανταγωνιστική, που θα παρέχει βιώσιμη κοινωνική ευημερία. Και καθόρισα ποιε πίστευα ότι είναι οι προσδοκίε των πολιτών για το μέλλον, για την ανάπτυξη, τη σταθερότητα, για τι δουλειέ, για την ευμάρεια. Όλοι ξέρουμε ότι περνάμε πολύ δύσκολου καιρού σήμερα. Και γι' αυτό ακόμα πιο σχετική γίνεται αυτή η πτυχή σήμερα που ανέφερα. Πρέπει να εργαστούμε για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερε δυνατότητε απασχόληση, επιφέροντα διαθροτικέ αλλαγέ. Και μάλιστα διότι το πεδίο για μακροοικονομικά κίνητρα έχει ε, εξαντληθεί, διότι τα δημοσιονομικά περνάνε μεγάλες πιέσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δυσκολίες. Για κάποιες χώρες δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική παρά η μείωση του βάρους του δημοσίου χρέους. Και αυτό είναι πάντα ένα βάρος που βαρύνει την επόμενη γενιά, που πληρώνει αυτά τα χρέη. Επίσης, είναι επιζήμιο για την εμπιστοσύνη και τις δυνατότητες ε, ανάπτυξης των κρατών μελών. Και επηρεάζει βέβαια αρνητικά και τις κοινωνίες. Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που έχουν μεγαλύτερη σημασία είναι αυτές που μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα να προσαρμοστούμε. Μακροπρόθεσμα η παραγωγικότητα θα εξαρτάται από καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Η κοινωνική συνέπεια της κρίσης ήδη είναι πολύ μεγάλη. Αυξάνονται δυστυχώς πολύ τα επίπεδα της ανεργίας και με απασχολεί τα μάλα αυτό. Κυρίως διότι έχει αυξηθεί πολύ η ανεργία των νέων. Τεράστια σπατάλη ταλέντου και ανθρώπινης ευημερία είναι αυτή. Και αυτό δεν μπορεί να το ανεχθεί η Ευρώπη, να το αντέξει η Ευρώπη. Αν ήμουν νέος Ισπανός, θα διερωτώ Γιατί έχουμε 20% ανεργία στην Ισπανία, ενώ στην Ολλανδία είναι 4% ή στην Αυστρία 5%. Τι πρόβλημα έχουν οι θεσμοί μας, οι πολιτικές μας, η λειτουργία της αγοράς εργασίας, γιατί έχουμε τόσο ψηλή ανεργία. Να μην μιλήσω για την ανεργία των νέων στην Ισπανία πάνω από 40%. Εδώ βλέπουμε πόσο χρειάζονται οι διάφορες διευθυντικές μεταρρυθμίσεις στα πλαίσια της ευέλικτης ασφάλειας και την προσπάθεια της δυνατότητας αυξήσεως της, των δυνατοτήτων απασχολήσεως των πολιτών μας. Θέλουμε να βελτιώσουμε λοιπόν την απασχολησιμότητα και την κοινωνική ευημερία στην Ευρώπη. Αυτός πρέπει θα είναι ο βασικός στόχος του έργου μας. Και γι' αυτό ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν προτεραιότητα συγκεκριμένες δράσεις που έχουν σαν στόχο ιδιαίτερος τους νέους που δεν ε, είναι μέσα σε πλαίσια απασχόλησης, κατάρτισης ή εκπαίδευσης. Και ο προκάτοχός μου, το, ο Λάς Λάντορ, ο συνάδελφός μου παρουσίασε το θέμα αυτό όσον αφορά τις πολιτικές που να ακολουθήσουμε για την απασχόληση. Ο Λάς Λάντορ. Λοιπόν, αξιότιμα μέλη. Θέλουμε να αναζωογονήσουμε την ανάπτυξη. Και η στρατηγική μας πρέπει να αποκαταστήσει την χρηματοπιστική και οικονομική σταθερότητα που έχει διαβρωθεί και διαβρώνει και στα θεμέλια της οικονομικής ανάπτυξης. Όσον αφορά την οικονομική σταθερότητα, μεσοπρόθεσμα, αυτό είναι κρισίμου σημασία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ έκανε πολλή δουλειά ήδη. Και συνεχίζει. Σε συνεργασία με τον συνάδελφό μου, τον Μισελ Μπαρνιέ, που είναι στη θέση του οδηγού, έχουμε αλλάξει ριζικά μαζί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το ρυθμιστικό και το υποπτικό πλαίσιο και την αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού πλαισίου της ε, Ευρώπης. Πολλά απομένουν να κάνουμε, αλλά ο χρηματοπιστωτικός τομέας πρέπει να παίξει τον οικονομικό και κοινωνικό του ρόλο σαν μια πηγή χρηματοδοτήσεως πραγματικής οικονομίας για την απασχόληση, για τις επιχειρήσεις και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα συμπεριλαμβάνει και το θέμα των τείχων προστασίας firewalls ή backstops. Όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα και το κρατικό χρέος για να ξεπεράσουμε την κρίση, η στρατηγική είχε διτή προσέγγιση αυτή που ακολουθήσαμε. Πρώτα απ' όλα δημιουργήσαμε διάφορα σημεία υποστήριξη χρηματοπιστωτικά για να εμποδίσουμε ε, την πιθανότητα χρεοκοπία των πολύ χρεωμένων κρατών μελών και να αποφύγουμε και επιμόλυνση στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη γενικότερα. Και δεύτερον, μαζί με αυτή την Επιτροπή αναλάβαμε μεγάλη μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ένωση, κάτι που θα βοηθήσει να μειώσει το ε, δημόσιο χρέος σε βιώσιμα επίπεδα και εξίσου σημαντικό να αποφύγει στο μέλλον επανάληψη τέτοιας κρίσης. Να πω μερικά λόγια για το πρώτο θέμα εκείνα τα σημεία στήριξη τα δημοσιονομικά. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο επέκρινε κάποιες πτυχές των μέσων της οικονομικής βοήθειας υπό συγκεκριμένου όρους, το EFSF και σύντομα το ESM, όσον αφορά τις θεσμικές πτυχές, δεν αποτελεί μυστικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τις ανησυχίες σας, τις μοιράζεται, η διακυβερνητική προσέγγιση ήταν χρονοβόρα, πολύ χρονοβόρα και δεν ήταν αρκετά αποτελεσματική και μόνο τώρα κάποιες από τις προτάσεις που κάναμε, ας πούμε εδώ και ένα χρόνο, μισή χρόνο, υλοποιούνται τώρα. Αναφέρομαι, παραδείγματο χάρη, στις εκκλήσεις που απευθύναμε εδώ και ένα χρόνο περίπου, τον Ιανουάριο, να ενισχυθεί η δυνατότητα δενεοδότησης του EFSF και να διευρυθεί και το πεδίο δραστηριοτήτων του μέσου αυτού, αυτό αποφασίστηκε τελικά μόνο στην Σύνοδο Κορυφής Ευρωζώνης το Οκτωβρίου. Και η τεχνική και νομική εφαρμογή θα πρέπει να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, στο Eurogroup. Τολμώ να πω ότι αν είχαμε αποφασίσει επ' αυτού εδώ και ένα χρόνο, Φερρυπίν, δεν θα ήμασταν σε τόσο βαθιά κρίση σήμερα, όπως είμαστε, δυστυχώς. Τι κάναμε μέχρι τώρα. Θέλω να εξασφαλίσουμε ότι η κοινοτική μέθοδος θα κρατήσει το ρόλο που έχει και ότι θα ενισχυθεί στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το EFSF και από το EFSM. Και σε δύο μέρες το πακέτο ανάπτυξης και διακυβερνήσεως θα υποβληθεί σε εσά. Θα περιέχει νομοθετικές προτάσεις για έναν κανονισμό που θα εντάξει την κοινοτική μέθοδο τα προγράμματα εποπτείας. Εκεί πραγματικά ανήκουν οι προτάσεις αντικατοπτρίζουν το εξή. Αποτελεσματική και αποδοτική εποπτεία δεν μπορεί να εφαρμοστεί μέσω διακυβερνητικής προσέγγισης με απαιτήσει περί ομοφωνίας. Συνεπώς αναγνωρίζεται και υπογραμμίζεται ότι μόνο ισχυροί θεσμοί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κοινοτική μέθοδος μπορούν να αποδώσουν και να πετύχουν τους στόχους Δηλαδή, υγιή οικονομική και δημοσιονομική εποπτεία. Αυτή είναι η βάση των προτάσεων των σημερινών, που βεβαίως εδράζονται επί του six-pack, που σύντομα θα τεθεί σε ισχύ. Τόσον αφορά τις ανησυχίες της Επιτροπής σας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν γέννη, σχετικά με την αποδοτικότητα του EFSF. Πιστεύω, παρόλα αυτά, ότι οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής Ευρωζώνης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, σημείωσαν σημαντική πρόοδο, δίκησαν σημαντική πρόοδο. Η ύψιστη προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι ταχεία και πιστή εφαρμογή των αποφασιστέντων. Για μόχλευση του EFSF προωθώντα το ESM, τη μόνιμο μηχανισμό στήριξη για να ενισχυθεί η, δυνατότητα, η δύναμη πυρό μα. και να ενισχυθεί μέσω ανακεφαλοποίηση ο χρηματοπιστωτικό τομέα και μέσω μεταρρύθμισης ε, στον τομέα το τραπεζικό. Και αυτό πρέπει να γίνει σύντομα. Η πρόληψη είναι ο δεύτερος κλάδος στρατηγικής μας. Πρώτη προτεραιότητα είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτά που συμφωνήθηκαν θα εφαρμοστούν επίση. Και Αναλαμβάνω πολύ σοβαρά αυτή την ευθύνη. Θα κάνω πλήρη χρήση όλων των νέων μέσων του Six Pack από την πρώτη μέρα κιόλα, που όπω επιβεβαιώθηκε θα είναι η 13η Δεκεμβρίου η πρώτη μέρα εφαρμογή. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε παραβίαση κανόνων κοινώ συμπεφωνημένων από κανένα κράτο μέλο. Αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει, διότι είδαμε με δραματικό τρόπο στην πραγματικότητα ότι αυτό συμβαίνει εις βάρος άλλων κρατών μελών, αυτή η παράβαση. Είναι εις βάρος άλλων κρατών μελών και των πολιτών. Είμαστε τόσο, υπάρχει τόσο μεγάλη εξάρτηση στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να σεβόμαστε τους κανόνες που έχουμε συμφωνήσει. Σύμφωνα βέβαια με τη δημοκρατική νομιμότητα που έχουν επικυρωθεί σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια αυτοί οι κανόνες. Λοιπόν κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σαν ένα μέρος της συμφωνίας για το Six Pack, θα θυμόσαστε, ότι είχαμε συμφωνήσει να σας παρέχουμε ανάλυση επιλογών για τα ευρωομόλογα ή ομόλογα σταθερότητας. Ε, παρουσιάσαμε πράσινη βίβλο επί των διαφόρων επιλογών για τα, αυτά τα ομόλογα σταθερότητας σήμερα μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, μετά από έντονες συζητήσεις και προετοιμασίε, εντατικέ μα συζητήσει και προετοιμασίε τι προηγούμενε ημέρε, ακόμα και μέχρι τα τελευταία λεπτά πριν υποβάλουμε τι προτάσει, και με την προοπτική να υποβάλουμε αυτά τα ομόλογα σταθερότητας, ίσως αυτά τα ομόλογα θα μπορέσουν να μειώσουν τα προβλήματα που έχουμε λόγω των κρατικών ομολόγων και του κρατικού χρέου. Βέβαια δεν, δεν έχουμε μία και μοναδική λύση που θα μας βγάλει, μία πανάκια που μας βγάλει από την κρίση. Πρέπει να κινηθούμε σε πολλαπλά μέτωπα και γι' αυτό οι σημερινές αποφάσεις πράγματι θα πρέπει να ειδωθούν σαν ένα συνολικό πακέτο που υπογραμμίζει βασικό στόχο την οικονομική ανάπτυξη και παρέχει συγκεκριμένες προτάσεις για να οδηγήσει σε αυτή τη βιώσιμη ανάπτυξη δημιουργία θέσεων απασχόληση που μπορεί να δημιουργηθούν αυτά και κάνοντα και διάφορα άλλα βήματα για την ενίσχυση τη οικονομική διακυβέρνηση, κυρίω στον τομέα στην περιοχή τη Ευρωζώνη. Και παράλληλα με αυτό, πώ θα ξεκινήσει η σοβαρή συζήτηση όσον αφορά αυτά τα ομόλογα σταθερότητα. Θα ήθελα λοιπόν σε ένα-δύο λεπτά που μου έχουν απομείνει να πω κάποια πράγματα για τις επιλογές που έχουμε όσον αφορά αυτά τα ομόλογα σταθερότητας. Έχουμε δώσει σχετική ανάλυση και τα δύο βασικά πορίσματα είναι τα εξή. Πρώτον, ναι, κοινώς εκδομένα τέτοια ομόλογα σταθερότητας πιθανότατα θα ήταν ουσιαστικά επωφελή, θα μείωναν και θα σταθεροποιούσαν το κόστος δανειοληψίας από πλευράς κρατών μελών διότι θα υπήρχε μεγαλύτερη αντίσταση στα σοκ όσον αφορά το χρηματοσυντικό τομέα και θα βελτιωνόταν και η αποδοτικότητα με την πάροδο του χρόνου της, ε, των αγορών. Αλλά σαν ομόλογα σταθερότητας, αυτά τα ομόλογα σταθερότητας και τα ευρωμόλογα θα μείωναν την ε, πειθαρχία των αγορών των ξεχωριστών κρατών μελών, αυτή η εισαγωγή τους θα είχε νόημα και θα ήταν πραγματιστική υπό τον όρο ότι η οικονομική διακυβέρνηση θα έπρεπε να ενισχυθεί ουσιαστικά κατά πολύ παράλληλα με την εισαγωγή αυτής της πιθανότητας εκδόσεως ομολόγων σταθερότητας. Το Six Pack ήδη είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και οι σημερινές προτάσεις ε, αντιπροσωπεύουν ένα περαιτέρω βήμα όμως ίσως θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις για να διευκολύνουμε μια ασφαλή εισαγωγή αυτών των ομολόγων σταθερότητας. Λοιπόν κυρίες και κύριοι θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι οι σημερινές προτάσεις βασίζονται επί των αποφάσεων τη Συνόδου Κορυφή τη Ευρωζώνη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου βασίζονται στην κοινή δουλειά που κάναμε όσον αφορά αυτό τη δέσμη μέτρων, το Six Pack και την ενίσχυση τη οικονομική διακυβέρνηση και παρέχουν ισορροπημένο αλλά αποφασιστικό δικό χάρτη για ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης που συνοδεύεται από διάφορες δυνατότητες για την εισαγωγή αυτών των ομολόγων σταθερότητας. Και εδώ θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστεύω να την υποστηρίζετε, θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών, όλων των πολιτών της Ευρώπης και να διαφυλάξει το κεκτημένο κυρίως της ενιαίας αγοράς και να εξασφαλίσει ότι οι αλλαγές όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση θα λάβουν χώρα διαφανώς, δημοκρατικός, κοινοτικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Όπως είπα, ο χρόνος πιέζει. Ένα λεπτό λοιπόν και θα είμαι αυστηρή. Οπότε αν δεν βιαστούν ε, οι πρώτοι ομιλητές, οι τελευταίοι δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν. Οπότε 10 δευτερόλεπτα παραπάνω να μιλήσει ο πρώτο σημαίνει 10 δευτερόλεπτα λιγότερα από τον τελευταίο και σοβαρό λόγο. Θα ακούσουμε τι ερωτήσει σε ομάδες των τριών για να έχει μετά και ο επίτροπο 6 λεπτά για να απαντήσει. Εάν δεν δουλεύει το σύστημα θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, τρει πρώτε ερωτήσει. Διόγκο Φέιο, Ελίζα Φερέιρα και Σιλβί Γκουλάρ. Διόγκο. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε Αλή Ρεν. Θα ήθελα να σας συγχαρώ καταρχάς για την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας καθώς επίσης και για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε για να λυθεί η κρίση του ευρώ. Επίσης θα ήθελα να σας συγχαρώ για το σύνολο του νομοθετικού πακέτου της δέσμης που καταθέσατε για να επέλθει ε, σταθερότητα και διακυβέρνηση. Με τα νέα σας καθήκοντα και τις νέες αρμοδιότητες τώρα θα μπορείτε να προεδρεύετε στο Eurogroup. Μιλήσατε για ένα νέο Ισπανό. Σε ποιο Ευρωπαίο νέο από οποιαδήποτε χώρα μπορείτε να εξηγήσετε τη στρατηγική σας για την ανάπτυξη. Τι συγκεκριμένα μέτρα θα τους λέγατε για τα λεγόμενα ομόλογα σταθερότητας. Αυτά τι είναι, σε ποιο βαθμό συνδυάζουν τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ανάπτυξη της οικονομίας. Πώς θα συνδυάζουν αυτά τα δύο. Και ένα τελευταίο, σας δείχνω την πειθαρχία των Πορτογάλων σε, ό,τι αφορά το χρόνο. Η κυρία Φερέιρα. Κύριε Επίτροπε, καλώς ορίσατε. Θα ήθελα να πω ότι και εσείς αναγνωρίζετε ότι έχει ε, αποτελματωθεί η οικονομία και η ανάπτυξη στις χώρες μας. Δεν υπάρχει όμως περιθώριο ελιγμών ούτε στο λεγόμενο six pack στη δέσμη των έξι οδηγιών ούτε στην ευρωπαϊκή στρατηγική. Έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις που έχουν διαταράξει την εμπιστοσύνη στη συνεργασία μας. Είχαμε συμφωνήσει κάτι για τους δείκτες ανταγωνιστικότητας, το οποίο ανετράπη. Εκτός από το μισθό και ε, το κόστος της εργασίας δεν έχετε άλλους δείκτες. Θετικά ή αρνητικά κατόφλια. Το μόνο που χρησιμοποιείτε είναι το μισθολογικό και το κόστος της εργασίας. Επίσης, δεν υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών. Μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό που είπε κάποιος Σουηδός υπουργό ότι η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρή οικονομία να είναι έτοιμες να βοηθήσουν να αναπτυχθεί η οικονομία σε όλη την Ευρώπη. Εγώ θα προτιμούσα αυτά να τα είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι ένας υπουργό Οικονομικών κάποιας χώρας. Αυτό ήταν 1,5 λεπτό. Οπότε υπερβάς θα μιλήσει μισό λεπτό η Σιλβί Κούλα. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε για την έκθεση για τα ευρωομόλογα που ζητούσε το Κοινοβούλιο, που επιθυμούσε και τηρήσατε το λόγο σας. Είναι αρκετά επιδέξιο να γίνει η πράσινη βίβλος γιατί πρέπει τα πράγματα να τα δούμε από την αρχή. Εγώ σας ρωτώ τις επόμενες εβδομάδες πώς θα βλέπετε η προθεσμία που έχετε ορίσει είναι πολύ μικρή, πολύ σφιχτή. Το Κοινοβούλιο θα κάνει βέβαια έκθεση πρωτοβουλία. Αλλά εσείς τι πιστεύετε, αρχές Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου αναμένετε να υπάρχει θέση και αν ναι, πού θέλετε να εστιάσετε την προσοχή του ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. That's your first three questions. Κύριε Επιτροπέ, αυτές είναι οι τρεις πρώτες ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Φέιο. Πρώτα απ' όλα για τα ευρωομόλογα. Πώς θα συνδυαστεί πειθαρχία με την σταθερότητα και πράγματι είναι σημαντική αυτή η ερώτηση γιατί ε, για να μιλήσουμε ειλικρινά εάν δεν έχουμε επαρκείς διαβεβαιώσεις δημοσιονομικής πειθαρχία. τα ευρωμόλογα εύκολα θα γίνουν και αυτά θα πέσουν στην κατηγορία junk σκουπιδιών. Οπότε, για να έχουμε ρεαλιστικά να έχουν νόημα τα ευρωομόλογα θα πρέπει ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την ε, οικονομική διοίκηση, διακυβέρνηση. Γι' αυτό η σημερινή πρόταση που βασίζεται στο άρθρο 136 όσον αφορά την επιτήρηση των εθνικών προπολογισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στην Ευρωζώνη και την ενισχυμένη επιτήρηση χωρών που αντιμετωπίζουν πιθανό κίνδυνο αστάθειας είναι τόσο σημαντικές. Είναι κρίσιμα βήματα προς μια όλο ένα πιο στενή η Οικονομική Ένωση, η οποία θα έχει τα απαραίτητα μέσα και βεβαίω επιτήρηση και τα μέσα για να επιβάλλει αυτή την επιτήρηση. Οπότε θα πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα πειθαρχία και σταθερότητα και όταν λέω σταθερότητα εννοώ σταθερότητα και από την έννοια της δημοσιονομικής πειθαρχίας και στις χρηματαγορές. Όσον αφορά το κέριο ερώτημά σα για το πώς θα εξηγήσουμε σε ένα νεαρό Ισπανό γιατί η Ισπανίδα, γιατί αντιμετωπίζει ε, ανεργία 46% που είναι το ποσό των άνεργων νέων στην Ισπανία οπωσδήποτε δεν είναι, είναι εύκολη η απάντηση και η διέξοδος αλλά ουσιαστικό είναι να ξεκινήσουμε τις μεταρρυθμίσεις τώρα. Και δράτω με τις ευκαιρίες να ενθαρρύνω την κυβέρνηση η οποία θα αναλάβει στην Ισπανία να αναλάβει τολμηρές μεταρρυθμίσεις για να μεταρρυθμίσει τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε προοπτικές των νεαρών Ισπανών να βελτιωθούν. Δεν είναι δίκαιο το ότι είναι τόσο χωρισμένη η αγορά εργασίας στην Ισπανία μεταξύ αυτών που είναι μέσα και αυτών που είναι στην απέξω με αποτέλεσμα το πολύ υψηλό ποσοστό που είναι πάνω από 20% συνολικά στη χώρα. Ε, πόση ώρα έχω ακόμα? Ε, έχω 6 λεπτά σύνολο. Τέλος πάντων. Συνήθως είμαι σύντομο. Η κυρία Φρέρα έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα, αλλά θέλω να δω κάποια στοιχεία, γιατί... Ε, δεν μίλησα με την κυρία Φεραίρα αλλά ανέμενα κάποιες ερωτήσεις. Όσον αφορά τους δείκτες. Αναμένουμε τα γραπτά σχόλια του Κοινοβουλίου για το τη μορφή αυτού του πίνακα βαθμολογία. η Κομισιόν δεν αναμένει μεγάλες αλλαγές δεδομένου του ότι Κοινοβούλιο και Συμβούλιο ε, έλαβαν μέρος στις τεχνικές συζητήσεις ούτως ή άλλως στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου που δεν είναι κάτι το πολύ συναρπαστικό βεβαίως αλλά ε, συχνά οι συζητήσεις αυτές είναι και μακροσκελείς και απαιτούν και αντοχή και σας ευχαριστώ. Όσον αφορά λοιπόν τη μορφή που θα έχει αυτός ο πίνακας βαθμολογίας, θα ήθελα να ευστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα στοιχεία τα οποία μας απασχόλησαν στις ε, τελευταίες φάσεις του τριμερούς ε, διαλόγου. Πρώτα απ' όλα σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε έναν δείκτη για την εξέλιξη της απασχόλησης. Δεύτερον, οι δείκτες ε, που σκοπεύουμε να που σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε θα έχουν ε, και την ανταγωνιστικότητα πλην των ε, τιμών για να έχουμε τα διάφορα μέτρα της παραγωγικότητας και έναν ευρύτερο δίκτυ του χρηματοπιστωτικού τομέα που σκοπεύαμε να έχουμε αλλά απαιτείται περαιτέρω τεχνική ανάλυση και σκοπεύουμε να το οριστικοποιήσουμε εντό του επομένου έτους και οπωσδήποτε εγκαίρως πριν το επόμενο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Με τις δε χώρες, ε, τις πλεονασματικές και τις ε, ελληματικές θα απαντήσω. Θα ασχοληθώ σε μια επόμενη ερώτηση. Απλά για αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκουλάρ. Να πω πως εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε την ε, πράσινη αυτή βίβλο ως ένα τμήμα ενός γενικότερου οράματος για το πώς να δημιουργήσουμε μια πραγματική οικονομική ένωση στην Ευρώπη. Γι' αυτό η σχέση μεταξύ του κανονισμού του 136 για ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας αφενός και αφετέρου τα ομόλογα αυτά σταθερότητας ε, είναι πράγματα τα οποία είναι εγγενώς συνδεδεμένα και γι' αυτό καλό όλα τα θεσμικά όργανα και εσάς του Κοινοβουλίου και τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω δισταγμούς και καθυστέρηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Οι επόμενες τρεις ερωτήσεις θα γίνουν από την Βίκη Φόρτ, τον Φιλίπ Λαμπέρτς και τον Γιούργεν Κλούτε, ο οποίος όμως απουσιάζει, οπότε θα είναι ο κύριος Χουντής. Βίκη, ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, όσοι είμαστε εκτός της Ευρωζώνης, ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη και η σταθερότητα της Ευρωζώνης για την δική μας ανάπτυξη. Αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ένα έλλειμμα του υπερπολογισμού πάνω από 8%, διπλάσιο από αυτό της Ευρωζώνης, πάνω από διπλάσιο από αυτό της Ιταλίας και παρόλα αυτά είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος καθαρός φορέας στον προπολογισμό της ε, Ένωσης που συμφωνήθηκε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και έχουμε συνεισφέρει ούτως ή άλλως κοντά στο 5% στις, διαδόσεις, στις διασώσεις μέσω δούνου του κτλ. Ε, μήπως είστε λίγο εγωιστές, κύριε Επίτροπε. Ο, Φιλίπ Λαμπέρτς. Κύριε Επίτροπε, θεωρώ πως ε, εμείς οι δύο συμφωνούμε πως δεν θα βγει η Ευρώπη από την κρίση χωρίς πολύ βαθύτερη δημοσιονομική ολοκλήρωση και πολιτική ολοκλήρωση, αλλά αυτό θα γίνει αν δεν αναγνωρίσουν οι πολίτε την νομοποίηση των αποφάσεων. Και αν διαβάσουμε το τι γίνεται, βλέπουμε πω η Κομισιόν παίρνει περισσότερε εξουσίε, έτσι ώστε να μπορεί κατ' ουσία να κατησχύει εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων χωρίς κανένα έλεγχο. Δηλαδή Συμβούλιο και Κομισιόν πίσω από κλειστέ ε, πόρτες θα μπορούν να έχουν τον τελευταίο λόγο έναντι εθνικών δημοκρατιών θα ήθελα να τονίσω πως αυτό το οποίο κάνει η Αγγέλα Μέρκελ όταν ζητάει ψηφοφορία από την Bundestag πριν έρθει στις Βρυξέλλες, λίγοι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες το κάνουν. Τα εθνικά κοινοβούλια ε, έχουν βγει ούτως ή άλλως από το παιχνίδι. Οπότε, τι βλέπουμε. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα βασικά τα οποία κάνει η Κομισιόν, δηλαδή ετήσια έρευνα ανάπτυξης, πολιετή αναπτυξης πολυετη στρατηγικη και αποφάσεις παρέμβασης κάτι σα πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ε, δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη έναντι της Ένωσης πρέπει να συζητηθούν και να εγκριθούν από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι τα ελάχιστα για να υπάρχει δημοκρατική νομιμότητα. Ε, δέκα δευτερόλεπτα από την επόμενη φορά. Κύριο Χουντή, για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, ζητάτε κι εσεί, δεν ξέρω αν είναι στα νέα σα καθήκοντα, γραπτέ εγγυήσει από ελληνικέ πολιτικέ δυνάμει και κόμματα της αντιπολίτευσης για την εφαρμογή της απόφασης της 26 Οκτωβρίου. Αυτό δεν προβλέπεται στην απόφαση. Τα κόμματα από τα οποία ζητάτε γραπτές δεσμεύσεις ήδη έχουν συμφωνήσει ότι θα ψηφίσουν τα απαράδεκτα μνημόνια και ό,τι θα επακολουθήσει χωρίς να το έχουν ερωτήσει, χωρίς να το έχουν μάθει. Επομένως αυτό που κάνετε είναι προσβολή στη δημοκρατία και προσβολή σε έναν ολόκληρο λαό. Σας ερωτώ λοιπόν, Πρώτον, υπάρχει άλλο προηγούμενο από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να ζητείτε τέτοια διαδικασία νομιμοποίησης αποφάσεων και από κόμματα της αντιπολίτευσης. Και δεύτερο, από ποιο άρθρο, ποια συνθήκης εσείς αντίλητε αυτό το δικαίωμα να παρεμβαίνετε στις εξελίξεις και στα εσωτερικά μιας χώρας, αναφέρετε αυτό στα καινούρια σας καθήκοντα. Thank uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτέ είναι οι ερωτήσει Αν είστε έτοιμος, απαντήστε. Ευχαριστώ, Σάρων. Όσον αφορά το ερώτημα της ε, κυρίας Φόρτ για το ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου τη στήριξη της Ευρωζώνης ε, για να ξεπεράσει την κρίση του δημοσίου χρέους. Δύο πράγματα θα πω. Πρώτα απ' όλα υπάρχει πολύ μεγάλη αλληλεξάρτηση και οπωσδήποτε είναι προς το εθνικό συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου να βοηθήσει την Ευρώπη να ξεπεράσει την κρίση αυτή του δημοσίου χρέους. Δεύτερον, Θέλω να εκφράσω την ε, γνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν ε, έχει κάποια σημασία, προς το Ενωμένο Βασίλειο για το ότι συνεισφέρει στην διατήρηση της ε, χρηματοοικονομικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη. Μια που αναφερθήκατε σε εγωισμό, δεν θα τοποθετηθώ από αυτού. Θα υπενθυμίσω πως ένας Βρετανός Πρωθυπουργός κάποια στιγμή είχε πει πως δεν υπάρχουν μόνιμες συμμαχίες, μόνο μόνιμα συμφέροντα. Και νομίζω πως αυτό καθοδηγεί την ε, πολιτική της, ε, της χώρας σας. Και όταν ο πατέρας μου, ο παππούς μου, ε, επίσης στον πόλεμο τον χειμερινό ξεκίνησε να υπερασπίζεται την Φιλανδία, ήδη ο κύριος Τσόρτσιλ είχε ξεκινήσει να μειώνει την στήριξη της του Ηνωμένου Βασιλείου προς τη Φιλανδία γιατί προέβλεπε μελλοντική συμμαχία με τη Σοβιετική Ένωση. Αυτά για το εθνικό ε, συμφέρον. Αλλά νομίζω πως ε, είναι προς το κοινό μας συμφέρον να είμαστε ισχυροί μαζί στην Ευρώπη. Προς τον κύριο Φιλίπ Λαμπέρτς που αναφέρθηκε στον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων και την δημοκρατική νομοποίηση. Συμφωνώ πλήρω και είναι κάτι το οποίο θέλει να κάνει η Κομισιόν και το συζητήσαμε με τον Αντιπρόεδρο σήμερα στην Επιτροπή των κ. Σεφκοβιτ, ε, στο σώμα των Επιτρόπων για το πώ θα εμπλακεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια παρά το ότι ε, Κατά κύριο λόγο πρόκειται για έργο των και ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων, αλλά θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τίνουμε μια χείρα προς τα εθνικά κοινοβούλια, έτσι ώστε στην αρχή αυτών των έξι οδηγιών και των υπολείπων μεταρρυθμίσεων να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε για να επιτύχουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Αναφερθήκατε στο ότι τα κοινοβούλια σε γενικές γραμμές δεν ε, εμπλέκονται. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκονται σοβαρά τα κοινοβούλια. Να υπενθυμίσω παραδείγματος χάρη την Δανία ή τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα τη Φιλανδία. Εκεί πέρα τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ένα σύστημα το οποίο είναι και αποτελεσματικό και έχει βεβαίως νομιμοποίηση. Σύστημα διαβούλευσης ε, για διάφορα ζητήματα που δεν οδηγεί σε καθυστερήσεις ε, της αποφάσης της Ένωσης, τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Και ελπίζω κάποια μεγαλύτερα κράτη-μέλη με πολύ ισχυρές ε, συνταγματικές ε, ρήτρε να μάθουν κάποια μαθήματα από κάποια μικρότερα κράτη-μέλη όπου η κοινοβουλευτική εποπτεία λειτουργεί και αποτελεσματικά και Σεβόμενη την ε, δημοκρατική νομοποίηση. Ο κύριος Χουντής έθεσε ένα ερώτημα που αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής όσον αφορά την ενθάρρυνση πολιτικών δυνάμεων να στηρίξουν πολιτικές που βοηθούν στην αποκατάσταση της σταθερότητας στην Ευρώπη. Ε, βλέπω πως ε, η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ευρύτερα έχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την Ελλάδα, ένα νόμισμα που έχει δύο πλευρές. Αφενός υπονοεί πως η Ελλάδα σέβεται τις συμφωνίες και εκπληρώνει τους όρους όπως έχουν οριστεί στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ε, αυτό είναι εφαγωνίζεστε, το έχουμε συμφωνήσει μαζί, πάκτα σουντ σερβάντα, οπότε αναμένουμε να ε, τηρηθούν τα συμφωνημένα και από την Ελλάδα. Και από την άλλη τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι έτοιμοι και διατεθειμένοι και στήριξαν την Ελλάδα ουσιαστικά σε οικονομικούς όρους και είναι πράγματι ένα συμβόλαιο, όπως είπαμε, κοινωνικό, ε, στο οποίο η εκπλήρωση των όρων είναι προαπαιτούμενο για να δοθεί βοήθεια στην Ελλάδα. Με βάση αυτό η Κομισιόν ενθάρρυνε ε, έναν ευρύ συνασπισμό εθνικής ενότητας και χαίρομαι για το ότι ε, έγινε μια τέτοια κυβέρνηση στην Ελλάδα και θέλουμε να συνεργαστούμε με την ελληνική κυβέρνηση, τη Βουλή των Ελλήνων, την κοινωνία και τον λαό για να μεταρρυθμιστεί η Ελλάδα και να αποκατασταθεί η οικονομική βιωσιμότητα της χώρας. Και έχουμε και πέντε δευτερόλεπτα. Ναι, αλλά είχατε ξεπεράσει κατά 27 την προηγούμενη φορά. Η επόμενη τριάδα ερωτήσεων. Η κυρία Κράτσα, ο Αντολίν Σάντσες Πρεσέδο και ο Βόρφ Κλίντς, ο οποίος εξαφανίστηκε, οπότε θα μιλήσει η Σοφή Νετφέλτη. Κυρία Κράτσα, παρακαλώ. Επίτροπε, ε, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω ήταν σχετικό με την ε, δημοκρατική νομιμοποίηση της νέας ε, δημοσιονομικής αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη, αλλά ήδη έχετε απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις. Γι' αυτό θα σας ρωτήσω ε, πώς βλέπετε, πώς αντιμετωπίζετε τις σκέψεις που διαμορφώνονται και τις προτάσεις που ακούγονται για έναν διαφορετικό και ενεργότερο, αποτελεσματικότερο καθαρότερο τρόπο, ε, ε, τρόπο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην αντιμετώπιση της κρίσης με νομισματικές μεθόδους παρέμβασης όπως το τύπομα χρήματος, ο θέσπις ορίου στα σπρέτς, η δανειοδότηση μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου των κρατών μελών. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Ο Αντολίν Σάντσες. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια, κύριε Αντιπρόεδρε. Ορισμένοι λέγουν ότι το πρόβλημα της κρίσης δεν είναι πρόβλημα των βασικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε των θεμελίων, αλλά της ασθενούς διακυβέρνησης και της σταθερότητας. Τώρα μιλάτε για ομόλογα σταθερότητας. Ε, Πηγαίνουν στην κατεύθυνση γιατί εξισορροπούν ε, την κατάσταση και αντιμετωπίζεται και το θέμα. Είπατε θα ρωτήσει ένας νεαρός Ισπανός τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση καινούρια για να αντιμετωπίσει την κρίση και τι μέτρα πρέπει να λάβει. Αλλά πρέπει να πούμε σε οποιοδήποτε νέο Ευρωπαίο τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη συνολικά για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Με την ίδια ταχύτητα με τις χώρες που έχουν τα προγράμματα, τα μνημόνια. Αυτά τα ευρωομόλογα πότε επιτέλους θα τα εφαρμόσετε. Τι χρονοδιάγραμμα έχετε γνωρίζοντας ότι είναι συμβατά, δεν χρειάζονται αναθεώρηση της συνθήκης, μπορούν από τώρα να εφαρμοστούν. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Ενετβέλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο συνάδελφος Φιλίπ Λαμπέρς για την δημοκρατική νομιμοποίηση. Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα χρειαζόμαστε βαθύτερες θεμελιώδεις αλλαγές στο σύστημα, περισσότερες εξουσίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και περισσότερη λογοδοσία ακόμα και ε, η δυνατότητα παρέτησης ατομικά κάποιων επιτρόπων. Σήμερα πώς θέλετε να ε, συμπεριλαμβάνονται άμεσα στις αποφάσεις ε, τα εθνικά κοινοβούλια, όχι να δίνουν εντολέ σε υπουργού έμεσα, αλλά να αναλαμβάνουν το μερίδιο τη ευθύνη, να είναι συνυπεύθυνα για πάρα πολύ αντιλαϊκά και αντιδημοφιλή μέτρα γιατί τώρα ερμηνεύονται όλα αυτά ως επιταγή των Βρυξελών. Αναθεώρηση της αγοράς εργασίας, των συντάξεων στις κάτω χώρες, ε, ε, τα θέματα των ε, στεγαστικών δανείων. Πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά, πώς θα ενέχονται τα Εθνικά Κοινοβούλια μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχετε λοιπόν την τρίτη τριάδα ερωτήσεων, οπότε θέλετε μπορείτε να απαντήσετε κύριε Επίτροπε. Μάλιστα, ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας ε, Κράτσα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και σέβεται τη συνθήκη, η οποία ορίζει σαφώς ότι η πρώτη προτεραιότητα και η σημαντικότερη στόχη της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι η σταθερότητα των τιμών και μετά μπορεί να υποστηρίζει και τους άλλους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο βαθμό που δεν διακυβεύεται ο πρώτος στόχος της σταθερότητας των τιμών. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ισχυρή ε, δρέωση και κατοχύρωση του ευρώ ως βασική αρχή και εγώ είμαι βαθύτατα προσιλωμένος σε αυτό και στο ρόλο έχει παίξει. Έχει παίξει ευρύτερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη διαχείριση ε, της ε, κρίσης, ένα ρόλο πυροσβεστικό, αλλά καταρχάς ε, εξασφάλισε με ακράδαντη αποφασιστικότητα τη σταθερότητα των τιμών και στη συνέχεια συνεισέφερε για να διαφυλαχθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των μηχανισμών. με μη συμβατικά μέτρα που ήταν τόσο απαραίτητα όσο και πρόσφορα. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Σάντσες Πρεσέδο για τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η νέα Ισπανική κυβέρνηση. Αναφέρθηκα εν μέρη σε αυτό προηγουμένως και σας παραπέμπω εκεί ε, για την αγορά εργασίας και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτόν τον καιρό εξετάζει και μελετά τις πολιτικές των κρατών μελών και εν ευθέτω χρόνο θα προβούμε και σε νέες συστάσεις. Θα ήθελα όμως εδώ να πω το εξής. Σα παραπέμπω στι συστάση του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν από λιγου μήνε βάσει πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου αποφασίστηκε από το Συμβούλιο και ισχύει πλήρω ε, είναι νομική σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωση προς την Ισπανία και είναι μια πολύ καλή αφετηρία. Δύο-τρία παραδείγματα μόνο. Πρώτον, το Συμβούλιο συνιστά η Ισπανία να λάβει δράση στην περίοδο 2011-2012 για να εφαρμόσει τη δημοσιονομική στρατηγική για τον προπολογισμό του 2011 και του 2012 και να διορθώσει ε, το σημερινό έλλειμμα το έτος 2013 σύμφωνα με τις συστάσεις της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για να φτάσει στους στόχους της ε, για το έλλειμμα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων και των ε, μηχανισμών που ισχύουν με αυστηρή εφαρμογή για τις περιφερειακές κυβερνήσεις. και ε, να αναλάβει και δράση σε περίπτωση που δεν είναι αναμενόμενη η εξέλιξη του προπολογισμού. Πολύ σημαντική αυτή η πρώτη σύσταση. Δεύτερον, προτείνεται αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού, να αυξηθεί το όριο συνταξιοδότησης και ε, τα συντάξιμα χρόνια που απαιτούνται καθώς αλλάζει το προσδόκιμο ζωής ε, και ε, θα πρέπει επίσης να προβλέπετε διαβίου εκπαίδευση και μάθηση για όλους τους εργαζομένους. Είναι και άλλες συζητάσεις, πέντε νομίζω, δεν θα επιμείνω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική εφετηρία όλα αυτά για τη νέα κυβέρνηση την ώρα που ετοιμάζει το κυβερνητικό πρόγραμμα. Βεβαίω ε, παραμένουμε πάντα σε διαρκεί ε, διαβουλεύσεις ε, με την Ισπανία. Έχουμε εταιρική σχέση και με την κυβέρνηση της χώρας και με τη Βουλή τη και προσβλέπω και στη μελλοντική πάρα πολύ στενή συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση που θα αναλάβει, όπως θα κάνουμε και με την απερχόμενη. Σε ό,τι αφορά τη θέση σε ισχύ των ομολόγων σταθερότητας, 8 Ιανουαρίου τελειώνει η περίοδος διαβούλευσης. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε λάβει τις απαντήσεις από τη διαβούλευση αυτή θα εξετάσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Η Σόφι Νετβέλτ ρώτησε πώς θα βάλουμε στην προσπάθεια αυτή και τα εθνικά κοινοβούλια, όχι ε, μόνο τυπικά και άτυπα και ουσιαστικά και πραγματικά. Όπως σας είπα, συμφωνώ απολύτως με το στόχο αυτό. Και έχει σημασία εδώ να τονίσουμε ότι και στους δύο κανονισμούς, υπό το άρθρο 136, τονίζουμε την ανάγκη της πάρα πολύ στενής συμμετοχής και συνεργασίας και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και επίσης διατρανώνουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να εμφανιστούμε ενώπιον των Εθνικών Κοινοβουλίων και να εξηγούμε τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν προκειμένου και να εξηγήσουμε και τις στάσεις για την εκτέλεση του προπολογισμού ή τα συγκεκριμένα μέτρα. Είμαι πρόθυμος να το πράξω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συλλογικό σώμα, εάν το επιθυμήσουν, ή το ζητήσουν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πραγματικά θέλω γνήσιο και ουσιαστικό διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Um, Ευχαριστώ πολύ. Γίνεται πολύ περίπλοκο ο κατάλογος, γιατί φεύγουν κάποιοι. Επόμενες τις ερωτήσεις. Κέ Σουίντον, Φιλίπ Λάμπερτς και Γκέι Μίτσολ. Και η πρώτη. Επίτροπε Ρεν, δεν σας ζηλεύω. Όλο και πιο δύσκολη γίνεται η δουλειά σας, κάθε μέρα πιο δύσκολη. Σήμερα περιγράφηκα από τις παρατηθές της ε, αγοράς τα, τα μέτρα της Bundestag για τα κρατικά ομόλογα της ε, Γερμανίας, γιατί πολλά ομόλογα γερμανικά δεν αγοράστηκαν. Ε, παρά την οικονομική ισχύ της Γερμανίας σε σχέση με όλα αυτά, το κόστος της χρηματοδότησης της Γερμανίας φαίνεται ότι γίνεται όλο και δεν απανηρώ. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει σε πολύ μεγάλη τιμή όσον αφορά τα άλλα ομόλογα, διότι η πώληση των γερμανικών ομολόγων δεν πήγε καλά και έπεσε 0,1% ε, έναντι του δολαρίου. 1% έναντι του δολαρίου. Οι κεφαλαγορές δεν, δεν έχουν εμπιστοσύνη. δεν θεωρούν τα μέτρα στην Ευρωζώνη είναι επαρκή. Μπορεί να σχολιάσετε αυτό το θέμα της χρηματοδότησης της Γερμανίας. Τι συνέπειες μπορεί να έχει σε άλλες οικονομίες και μελλοντικά σχόλια τι θα γίνει στο μέλλον όσον αφορά την κοινή χρηματοδότηση των χρεών μέσω της εκδόσεως αυτών των ομολόγων σταθερότητα. Ο Φιλίπ, θα μιλήσω για την έκθεση για την ετήσια ανάπτυξη και να πω ότι περιέχει καλά στοιχεία όσον αφορά τη φορολόγηση, διότι έχει ενισχυθεί ε, αυτός ο τομέας έναντι άλλων ετών. Είδαμε αναφορές στην αύξηση της στόχια και ότι χρειάζονται διάφορα οικονομικά μέτρα, ώστε να μην υπάρχουν ε, αρνητικές συνέπειε ανακατανομή. Αυτό έχετε καθυστερημένα όσον αφορά τη φορολόγηση. Λείπει εξοπιστία από το έγγραφο, κοιτάζει τα πράγματα από τη μεριά των επενδύσεων και η στρατηγική σα στην ανάπτυξη εξασφαλίζει ότι θα καταναλώνουμε περισσότερο και θα πουλάμε περισσότερο. Υπάρχει μεγαλύτερο εμπόριο και δεν τονίζεται επαρκώ η πλευρά των επενδύσεων που πιστεύω ότι είναι στην προτεραιότητα σήμερα, ώστε η οικόνομη μα να γίνεται αποδοτική όσον αφορά την ενέργεια και, και του πόρου γενικότερα. Και εκεί που θα μπορούσαμε να επιφέρουμε βελτιώσει. Ευχαριστώ, οκ. Okay. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Η καλή διακυβέρνηση είναι απαραίτητη. Αλλά οι κυβερνήσει θα πρέπει να διακυβερνήσουν. Με εξέπληξαν αυτά που είπατε για τον ε, νέο Ισπανό και για τους νέους Ιρλανδούς και Ιρλανδές που είναι άνεργοι. Ε, ε, είναι άνεργοι. Δεν ήταν το Νητή είπε ότι αν υπήρχε σύμφωνο ανάπτυξη για ανάπτυξη στην Ασία και δημιουργία υποδομών στη Δύση, θα αναπτυσσόταν πολύ ταχύτερα η οικονομία και 25 με 50 εκατομμύρια θέσει απασχόληση θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη να προωθήσει αυτό το στόχο του Δούνου του, ε, το υποστηρίζετε, πότε θα δημιουργηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας. Έχουμε κολλήσει μήπως στους κανόνες, είμαστε τόσο κοντά στο δάσο που δεν βλέπουμε τα δέντρα. Τι συμβαίνει με αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Νομίζω ότι ακούσαμε τρεις ερωτήσεις. Έχω χάσει το μέτρημα κάπου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. το ερώτημα της ΚΕΙ. Για τις εξελίξεις όσον αφορά τα γερμανικά ομόλογα. δεν σχολιάζουμε καθημερινά τις, τα γεγονότα της αγοράς. Αυτό δεν είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθούμε να αποφύγουμε βραχυπρόθεσμα καθημερινά σχόλια. Όσον αφορά τον τομέα, γνωρίζουμε όλοι ότι η παρούσα κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι άκρως ανησυχητική, χειροτερεύει καθημερινά και αυτό υπογραμμίζει τη σημασία που έχει πρώτα απ' όλα να εφαρμόσουμε με αποφασιστικότητα τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής, των συνόδων κορυφής του Οκτωβρίου όσον αφορά τη διαφύλαξη της χρηματοστητικής σταθερότητας, ενισχύοντας τους τείχους προστασίας, τα τείχη προστασίας, τα οικονομικά και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να πάρουν σημαντικά ε, μέτρα αποφασιστικά για την αλλαγή την διαθροτική όχι μόνο πρέπει να ενθαρρύνουμε βραχυπρόθεσμες αποφάσεις για την αποκατάσταση εμπιστοσύνης, αλλά χρειάζεται και συγκεκριμένο μελλοντικό όραμα για να ισχυροποιηθεί η οικονομική μας ένωση και να γίνει στενότερη, όπου είναι αποτελεσματική η δημοσιονομική εποπτεία και οι μαϊκροοικονομικές ισορροπίες εκ των προτέρων ε, διορθώνονται. Αυτή είναι η προσέγγιση και αυτό υπογραμμίζει μόνο τη σημασία, την ύψιστη σημασία που έχει συντονισμένη και αποφασιστική δράση τώρα, σαν Ευρώπη. Ο Φιλίπ Λαμπέρτς αναφέρθηκε στις συνέπειες της ανακατανομής του πλούτου, τονίζοντας περισσότερο την έκθεση, την ετήσια για την ανάπτυξη θα πρέπει να το δείτε αυτό σαν σοβαρή απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακούει τους πράσινους, όλες τις πολιτικές οικογένειες και λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα σχόλιά σας και τα εφαρμόζει στο βαθμό των αρμοδιοτήτων μας στους τομείς αυτούς. Όσον αφορά την αποδοτικότητα των πόρων, χάρη στους συναδέλφους μου, Ποτότσνικ και η Χέρεκαρτ έχουμε ενισχύσει ουσιαστικά την αποδοτικότητα των πόρων για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Εμπεριέχεται και τονίζεται αυτό το στοιχείο. Εγώ δεν βλέπω όμως πρόβλημα, αντιθέτως να ενισχυθεί περαιτέρω αυτή η πτυχή και να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις ούτως ώστε οι οικονομίες μας να γίνουν πιο αποδοτικές όσον αφορά τους πόρους διότι όλοι ασχολούμεθα με την κρίση και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε τις οικονομίες μας πιο αποδοτικές όσον αφορά τους πόρους και αυτό μέσω μακροπρόθεσμα είναι απαραίτητο για να έχουμε βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ευημερία. Ο κύριος Μίτσελ αναφέρθηκε στην ε, διακυβέρνηση και τις κυβερνήσεις και κάποιες συστάσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό μου θύμισε κάποια πράγματα, διότι εμπεριέχονται στι συστάσεις των G20. Οι αποφάσεις ή δεσμεύσεις των G20 το θυμίζουν αυτό για την επανεξισορρόπηση της παγκόσμιας ανάπτυξης και τη διατήρηση οικονομικής ανάκαμψης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλες τις οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης και τη Ευρωπαϊκή οικονομία και των οικονομιών των κρατών μελών. Αυτή είναι η θέση που εκφράστηκε στο πλαίσιο των G20 για την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτό το θέμα συνέβαλε στις συζητήσεις και είδαμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε πολλά όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη αν καταφέρουμε να έχουμε πιο ισορροπημένη παγκόσμια ανάπτυξη και ένα καλύτερο μοντέλο για την ανάπτυξη. Αν απλουστεύσω τα πράγματα, μπορώ από τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η Ευρώπη πρέπει να λύσει τα του οίκου της αμέσως, τα προβλήματά της. Αυτό είναι που συζητούμε σήμερα. Και σήμερα και αύριο πάνω σε αυτόν τον άξονα κινούμαστε. Δεύτερον, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να λύσουν τα προβλήματά τους όσον αφορά το τεράστιο οικονομικό τους έλλειμμα και το βάρος του χρέους και σχετικά με αυτό είναι ατυχέστατο το ότι η Επιτροπή Εμπορίου δεν πέτυχε συμφωνία επί του σημαντικότατου αυτού στόχου. Και τρίτον, η Κίνα είναι από τις πιο μεγάλες οικονομίες που έχει πλεόνασμα και θα πρέπει να εξισορροπήσει το δικό της μοντέλο ανάπτυξης και να το στρέψει προς κατανάλωση και να ενισχύσει την ιδιωτική κατανάλωση που είναι βασικό στόχος του 12ου πενταετούς σχεδίου της Κίνας που είναι το εγχειρίδιο αν θέλετε της κινέζικης οικονομίας και αυτό σχετίζεται με την επανεξισορρόπηση των ισοτιμιών που θα οδηγήσουν σε παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Συμφωνώ πολύ με αυτές τις ιδέες και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούμε με τις ε, δεσμεύσεις που αναλάβαμε στα πλαίσια των ε, συζητήσεων των G20. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενοι τρεις, Λενάρντο Ντομένιτσι, Σιλβί Γκουλάρ για την Άλτε και Μάριαν Τάισεν για το ΕΛΚ. Λενάρντο. Κύριε Επίτροπε, λέτε ότι δεν χρειάζεται να σχολιάζεστε, να σχολιάζετε καθημερινά τις ειδήσει. Όμως το πρόβλημα είναι ότι σήμερα η κατάσταση επιδεινώνεται. Ε, καταλαβαίνετε το ποδόσφαιρο. Πάντα παίζεται άμυνα, αυτοί παίζουν άμυνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παίξει επίθεση το πρωί και δεν είναι σίγουρο τι γίνεται στο κέντρο. Ποια είναι η διασύνδεση με την... από την παρούσα κατάσταση με τις προοπτικές. Ποια είναι τα μέτρα που είναι σημαντικά που θα πρέπει να θετηθούν. Η επαναπρόθεση τη κοινοτική μεθόδου είναι ένα στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να προωθήσει σαν στόχο πολιτικό και θέλετε εσεί να το προωθήσετε ή πιστεύετε να το αναθέσετε σε διάφορου τεχνοκράτε. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο από τον Chief Economic Analyst της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Σιλβί. Ναι, κύριε Επίτροπε, σύντομα, γιατί χρειάστηκε να φύγει ο κύριος Κλίντς. Δεν είναι απλή ερώτηση, είναι όμως σύντομη. Τι γίνεται με τα διάφορα σχέδια και μορφές που παίρνει το Ταμείο Σταθερότητας. Αυτά που ακούω είναι πολύ αποκαρδιωτικά. Ε, κάναμε προσπάθειες, αποφάσεις είχαμε εθνικών κοινοβουλίων, δεν προχωρεί. Άλλες χώρες αποκλείουν ε, τα ευρωομόλογα, κάποιες άλλες ε, την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε κανένα μπούσουλα που πηγαίνουμε και πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ Μαριάν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, να σας συγχαρώ για τα νέα σας καθήκοντα και χαίρομαι για το ότι πράσινη βίβλος για τα ευρωομόλογα θα δημιουργήσει συζητήσεις στο πολιτικό επίπεδο, αλλά Βεβαίω θα πρέπει πριν υλοποιηθούν αυτά να υπάρξει μια οικονομική ε, σοβαρή διακυβέρνηση. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι οι δύο προτάσεις νόμου, πρόταση κανονισμού που ε, υποβλήθηκε σήμερα εκεί πέρα αναμένεται μια χαλαρή τοποθέτηση των κρατών μελών για να εφαρμοστεί γρήγορα και δεύτερον όσον αφορά τα ευρωομόλογα. Μήπως δεν θα ήταν καλό να λάβουμε μία απόφαση η οποία θα τα συνδέσει με κάποια έργα και βεβαίως αυτό για να στείλει και μήνυμα στις αγορές αλλά και να ενθαρρύνει και τα κράτη-μέλη για να βάλουν γρηγορότερα τάξη στα του οίκου τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να σας προειδοποιήσω, οι επόμενοι μιλητές θα είναι οι και εκεί πέρα τελειώνει ο κατάλογός μου, οπότε μπορείτε να μου πείτε ποιος θα ακολουθήσει. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το ερώτημα του κύριου Ντομένιτσι, να ξεκαθαρίσω το τι είπα. Δεν θέλουμε εμείς να σχολιάζουμε κάθε μέρα τις εξελίξεις στην αγορά. Ε, αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα κάνουμε σχολιασμό. Πράγματι θα το κάνουμε. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα δουλεύουμε για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ρωτήσατε ποια είναι η συνταγή μας θέλετε, για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έρευνα ανάπτυξης και η ετήσια έρευνα ανάπτυξης μαζί με το πακέτο ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης που βασίζεται στην ε, κοινοτική μέθοδο και με μια σοβαρή συζήτηση για την ε, πιθανή εισαγωγή ομολόγων σταθερότητας είναι θεωρώ εγώ μια αρκετά πιστική συνταγή και προς τα εκεί πρέπει να εργαστούμε. Μάλιστα σημερινό πακέτο δεν είναι κατενάτσιο, είναι ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, ε, επιθετικό περισσότερο που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρώπη. Και αυτό αναμένουμε από τα κράτη-μέλη στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μετά αναμένω να εγκρίνουν τις πολιτικές κατευθύνσεις της ε, σημερινής ε, ετήσιας ε, έρευνας ανάπτυξης και το υπόλοιπο πακέτο. Μάλιστα, έρχομαι έτσι στην απάντηση της κυρίας Γκουλάρ για αυτό το οποίο, όπως πολύ ωραία περιγράψατε, τις διάφορες ενσαρκώσεις των ε, ταμείων σταθερότητας. Πράγματι έχουν διάφορες μορφές. Είναι κάτι το οποίο συνεχώς εξελίσσεται και να σας εξηγήσω εγώ πώς το βλέπω. Να σας εξηγήσω το βασικό σκεπτικό πίσω από το σημερινό πακέτο. Ο δικός μας ε, χάρτης όσον αφορά την διασφάλιση της ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ε, έχει τρία κυρία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, σχολίασα ήδη τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν θέλω να επαναλάβω τις απόψεις μου. Παίζει και εξεκολουθεί να παίζει έναν ε, πολύ σημαντικό ρόλο, ε, πυροσβεστικό θα έλεγα. Δεύτερον, πρέπει να συμπληρωθεί η τεχνική εργασία όσον αφορά τη μόχλευση του EFSF για να αυξηθεί η δύναμη πυρός του ταμείου αυτού και αυτό πρέπει να γίνει μέχρι την ερχόμενη Τρίτη, το Eurogroup, γιατί η κατάσταση καθημερινά είναι πλέον εξαιρετικά κρίσιμη. Επιπλέον πρέπει να εγκρίνουμε νωρίτερα την ε, συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που βασίζεται σε κεφάλαιο καταβληθέν ε, και καταβλητέο το οποίο πλέον το καθιστά ένα πολύ πιο εύρωστο ε, οικονομικά μέσο από το EFSF. Οπότε αν έχουμε ένα μοχλευμένο ε, EFSF και εάν ε, φέρουμε πιο, αν δημιουργήσουμε πιο νωρίς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το ESM, τότε έχουμε ένα πολύ σοβαρότερο πακέτο για να περιορίσουμε, αν θέλετε, την μετάδοση της κρίσης. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό. Το τρίτο στοιχείο ε, είναι και επαναλαμβάνω σχεδίζεται με την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και έρχομαι εδώ στο ερώτημα της κυρίας Τάισεν ε, την πιθανή εισαγωγή κάποιας, ε, κάποιου είδους ομολόγων σταθερότητας κατά τρόπον ώστε να ενισχυθεί και η δημοσιονομική πειθαρχία και η σταθερότητα στην Ευρώπη. Χρειάζεται λοιπόν, όπως είπα, ένας οδικός χάρτης και πιστεύω πως ε, η σημερινή έρευνα που δημοσίευσαμε και τα υπόλοιπα στοιχεία, η πράσινη βίβλος για τα ομόλογα, οι δύο κανονισμοί για την οικονομική διακυβέρνηση μας δίνουν έναν οδικό χάρτη και για άμεσες λύσεις στην ε, κρίση η οποία μένετε, αλλά και για να διασφαλίσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να δημιουργήσουμε τις βάσεις ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Δύο ακόμα ε, παρεμβάσεις θα ακούσουμε. Περβάνο Μπερές και Παύλο Κατοπίν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, επιμείνατε επί του γεγονότος ότι θα πρέπει να γίνει όλη η προσπάθεια που και να βασίζεται επί της διαστάσεως της δημοκρατικής νομιμότητας. Άρα θα ξαναενστερνιστείτε τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Πριν το Συμβούλιο του Αρινό θεωρούσατε ότι σχεδόν ήταν νομοθετικές οι προτάσεις. Προτάσεις, που, θέσεις που θα άλλαζαν την ετήσια ε, εξέταση της ανάπτυξης και θα αναγνώριζαν ότι η εξέταση όλο αυτό το εγχείρωμα δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα του, αντι... του αντικειμένου που αποκαλείται έγγραφο προσανατολισμού. Μπορείτε να επικρίνετε κάθε κάτω μέλος που θα σας έστελνε ένα πρόγραμμα εθνικών μεταρρυθμίσεων που δεν θα αποτελούσε αντικείμενο εξέτασης εμβριθούς από τα εθνικά κοινοβούλια, από το συγκεκριμένο μάλλον εθνικό κοινοβούλιο του συγκεκριμένου κράτους. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Είπατε ότι αν ήσασταν νέος Ισπανός θα ε, σας προβλημάτιζε γιατί είναι τόσο μεγάλη ενεργεία. Και μένα με ανησυχεί αυτό ως Ισπανό και ως νέο γιατί ακόμα θεωρώ τον εαυτό μου νέο. Αυτό που είπατε ήδη ε, έχει εμφανιστεί στον Ισπανικό ψηφιακό τύπο. Από τώρα. Μιλήσατε για την ανάγκη αναθεώρησης αγοράς εργασίας στην Ισπανία και συμφωνώ. Είναι δύσκολη ερώτηση. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που συνιστάτε στη μελλοντική ισπανική κυβέρνηση ακριβώς για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέλος των ερωτήσεων εδώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να ελέγξω αν ενέκρινε το ψήφισμα ε, το Κοινοβούλιο για την ετήσια επισκόπηση για το 2011. Γιατί το περίμενα πολύ καιρό και λέγαμε πως μου είχε ξεφύγει. Όχι, δεν μου ξέφυγε. Ουσιαστικά γιατί δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα. Αλλά Πραγματικά μου λείπει γιατί ε, στην ουσία θέλω να έχω και το ψήφισμά σας αλλά και τις απόψεις σας για να ε, τα ενσωματώσουμε στις δικές μας πολιτικές αυτά που λέτε εσείς και που είναι πολύτιμα για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση. Λοιπόν, ας κάνουμε βαθιά συζήτηση για αυτό το θέμα και πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε πολύ εντατική και έντονη ανταλλαγή απόψεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσβλέπω στο ψήφισμά σας για το 2012 πλέον για να υπάρχει δημοκρατική νομιμότητα <coughs> ως έκφραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεδομένη. Αναφερθήκατε στα εθνικά ε, προγράμματα μεταρρυθμίσεων και αν περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκριθούν και να υιοθετηθούν από τα εθνικά κοινοβούλια. Έχουμε την άποψη ότι όλα τα βασικά έγγραφα και όλες οι βασικές αποφάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίζονται από ε, τα πολιτικά όργανα που έχουν δημοκρατική νομιμότητα. Δηλαδή για οποιαδήποτε στρατηγική απόφαση, ε, αυτή είναι τα εθνικά κοινοβούλια, όπως είναι τα εθνικά προγράμματα των μεταρρυθμίσεων. Αναμένουμε λοιπόν τα προγράμματα αυτά, τα μεταρρυθμιστικά των κρατών, να εγκριθούν από τα εθνικά κοινοβούλια και αυτό είναι αρμοδιότητα και καθήκον των εκάστοτε κυβερνήσεων. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω και να υπογραμμίσω αυτό που είπα προηγουμένω απαντώντα στην κυρία Νιτβέλτ. Βεβαίω και θέλουμε να έχουμε επικοδομητικό διάλογο με τα Εθνικά Κοινοβούλια και η πρόθεσή μου, όπω και του Αντιπροέδρου Σεύκοβιτς ε, και εξ ονόματος ε, του Συνόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι να προσκαλέσουμε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων ας πούμε τους προέδρους των Επιτροπών Προϋπολογισμού, των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για να κάνουμε ε, διαβουλεύσεις και ε, ένα είδος εργαστηρίου ας πούμε, για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην οικονομική διακυβέρνηση. Και βεβαίως με μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων προς το στόχο αυτό. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας για την ανεργία στην Ισπανία και τις μεταρρυθμίσεις ε, και της αγοράς εργασίας, θα σας έλεγα ότι προσωπικά Θα έμπαινα στον πειρασμό να συζητήσω και συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά αυτό το καιρό το επεξεργαζόμαστε το, αυτό το θέμα. σας είπα, είμαστε στη συνέχεια των συστάσεων, είμαστε σε διάλογο με τη δημόσια διοίκηση και τι υπηρεσίε τη χώρα, την απερχόμενη όσο και τη μελλοντική κυβέρνηση. Γι' αυτό προτιμώ να μην επεκταθώ, να μην μπω σε πολλέ λεπτομέρειε. Παρόλο που θα το ήθελα. Αλλά θα πρέπει ε, να πούμε ότι το βασικό ζήτημα είναι να μειωθεί ο διτός χαρακτήρας της ισπανικής οικονομίας. Και αυτό είναι ένας στόχος που πρέπει να αντιμετωπίσει η ισπανική κυβέρνηση. Διότι τέτοια ανεργία, 20% συνολικά και πάνω από 40% ανεργία των νέων, είναι απλούστατα κάτι το αφόρητο και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση για να μειωθεί αυτός ο υψηλός δείξης ανεργίας στην Ισπανία. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που ήρθατε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας μαζί μας. Βεβαίως η κυρία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μας δώσατε ειλικρινές, ειλικρινείς απαντήσεις ε, και ε, ευθείε και μερικές άλλες ε, κομψές. Προσβλέπω σε επόμενη συνάντησή μας. Ελπίζω να μας φέρετε καλά νέα την εφαρμογή της νομοθεσίας που μόλις εγκρίναμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Okay, Λοιπόν, συνεχίζουμε, πιέζει ο χρόνος. Καθίστε και πάλι σας παρακαλώ, γιατί έχουμε και δεύτερη ακρόαση που ε, προκλήθη από τον ελαφρύ ανασχηματισμό ε, των χαρτοφυλακίων Τον επιτρόπων. Όπως ακούσατε, ο Επίτροπος ε, Παρόσο αποφάσισε να αναθέσει ε, τη Eurostat στον Επίτροπο κύριο Σεμετά για να είναι ανεξάρτητη συλλογή στατιστικών στοιχείων και καλωσορίζουμε τον Επίτροπο κύριο Σεμετά για να μας μιλήσει για τη Eurostat, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και θα συνεχίσουμε με τη διαδικασία των ερωταποκρίσεων έχουν φύγει και ορισμένοι που θα έκαναν ερωτήσεις. Αν έχετε τίποτα να προσθέσετε ή κάποιος άλλος ε, θέλει το λόγο να ζητήσει γιατί κρατάω κατάλογο. Ε, θα δώσω το λόγο πρώτα στον Επίτροπο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με γνωρίζετε ως Επίτροπο Φορολογίας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τα φορολογικά γιατί βγήκε η αιτήσια έρευνα για την ανάπτυξη και περιέχει και ένα τμήμα ε, για τη φορολογία που αποτελεί πλέον ε, τακτικό μέρος στο Ευρωπαϊκό Εξωμήνου. Αλλά σήμερα θα μιλήσω για τα στατιστικά στοιχεία. Ο πρόεδρος Μπαρόσο μου έδωσε την ευθύνη της Eurostat. Είναι πεπισμένος πως έτσι θα ενισχύσουμε την ανεξαρτησία και την ε, αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων για να οδηγηθούμε σε καλύτερη εφαρμογή της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία είναι βεβαίως προαπαιτούμενο για να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις και από τους πολιτικούς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και άρα είναι ουσιαστική σημασία για τη δημοκρατία. Τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία είναι καλή ποιότητα. Όμω, επί τη βάση τη προσωπική μου εμπειρία ω επικεφαλή Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως τα στατιστικά στοιχεία είναι τόσο αξιόπιστα όσο τα θεωρεί το κοινό. Οι στατιστικοί φορείς δεν πρέπει μόνο να δρούν ανεξάρτητα αλλά και να φαίνονται ε, ανεξάρτητες και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε καιρούς ταραχώδης ε, όταν τα συναισθήματα παίζουν σημαντικότερο ρόλο από τα στοιχεία και όπου η αξιοπιστία ή η έλλειψη αυτής έχει παγκόσμιες συνέπειες. Οπότε η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της ανεξαρτησίας θα είναι η φιλοδοξία μου και έχω την πρόθεση με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αντιμετωπίσω αυτές τις προκλήσεις τους επόμενους μήνες. Η διακυβέρνηση στον τομέα των στατιστικών στοιχείων έχει ενισχυθεί στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Καλωσορίζω ιδιαίτερα την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Κώδικα Συμπεριφοράς καθώς και του Συμβουλευτικού Συμβουλίου. Θεωρώ όμως πως χρειάζονται ακόμα κάποιες ενισχύσεις για να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας παγκοσμίας τάξεως σύστημα ένα τάξιο σύστημα για τα στατιστικά στοιχεία. Τα απαραίτητα στοιχεία είναι πρώτα απ' όλα να διασφαλιστεί η επαγγελματική ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Δεύτερον, να υπάρξει αποτελεσματικό συντονισμό των εθνικών στατιστικών συστημάτων και τέλος οι εθνικές κυβερνήσει να γίνουν ρητά συνυπεύθυνε για την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων. Όλες αυτές οι πτυχές πρέπει να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα συμπεριληφθούν σε μια μελλοντική πρόταση τροποποίησης του κανονισμού για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία. Θα επιταχύνω το έργο αυτό για να συμποβάλλω αρχές του επομένου έτους μια νομοθετική πρόταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη καταστήσει σαφές πως αποδίδει μεγάλη σημασία στην επαγγελματική αξιοπιστία των στατιστικών αρχών σε εθνικό επίπεδο και την ανάγκη να προστατευθούν από πολιτικές παρεμβάσεις. Το καθεστώς του Διευθυντή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ήταν αντικείμενο πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει εισαχθεί επιτυχώς στο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης που υιοθετήθηκε πρόσφατα η Κομισιόν. Θα αναπτύξει αυτή την ιδέα στην πρόταση που θα υποβάλει ένα νέο μέσο επίσης θα δημιουργηθεί οι δεσμεύσεις για την εμπιστοσύνη στα στατιστικά στοιχεία θα είναι πολιτικές δηλώσεις που θα τονίζουν την εμπιστοσύνη των κυβερνήσεων στα ε, στοιχεία αυτά και στον κώδικα συμπεριφοράς θα τονίζουν ιδιαίτερα την ανεξαρτησία των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών από πολιτική επιρροή. Αναμένω τέτοιες δεσμεύσεις να γίνουν από όλες τις κυβερνήσεις. Θα είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι πως η Ένωση συνολικά δίνει μεγάλο βάρος στην αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων ε, όπως αυτά παράγονται από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Επίσης, θεωρώ πως η Κομισιόν πρέπει να λάβει τον ηγετικό ρόλο εδώ πέρα. Πρέπει στη Eurostat να εφαρμόσουμε τις αρχές που συστήνουμε στα κράτη-μέλη ένα καλό παράδειγμα έχει ήδη δημιουργηθεί. Με απόφαση του Προέδρου Μπαρόσο η Eurostat έγινε ανεξάρτητη από τους χρήστες των δεδομένων της, τους αναλυτές και αυτούς που χαράσουν την πολιτική εντός της Κομισιόν. Ο κίνδυνος πολιτικής παρέμβασης έχει μειωθεί κατά πολύ. Ένα άλλο σημαντικό βήμα πρέπει να ακολουθήσει. Σύντομα η Κομισιόν θα αναθεωρήσει την πολιτική της απόφαση για τον ρόλο της Eurostat με, ρόλ, με στόχο να ενισχυθεί η πολιτική ανεξαρτησία και ο σωρινιστικό ρόλο τη Eurostat. Η ανεξαρτησία του Γενικού Διευθυντή τη Eurostat από εξωτερική παρέμβαση κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα τονιστεί ιδιαίτερα. Επιπλέον, σκοπεύω να υπάρξουν να υπάρξει ένας νέος τρόπος λειτουργίας και εργασίας της ε, Κομισιόν που θα έχει και πάλι τη μορφή μιας δέσμευσης για την ανεξαρτησία της Eurostat. Πέρα από αυτή την ενισχυμένη στατιστική διαχείριση σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τα εθνικά στατιστικά στοιχεία. Θα φροντίσω η Eurostat να χρησιμοποιήσει πλήρως όλες τις, τις εξουσίες, οι ελεγκτικές εξουσίες που της έδωσε ο νομοθέτης πέρσι, αλλά και οι ε, αρμοδιότητες έρευνας που υπάρχουν στο εξαπλό πακέτο. Η Eurostat θα εξετάσει όλα τα δεδομένα πηγές σε περιπτώσεις σημαντικού κινδύνου και έρευνες εις βάθος θα διεξάγονται εάν υπάρχει υποψία ε, λαθροχειρίας στα δεδομένα και θα επιβάλλονται και πρόστιμα. Κατά την άποψή μου, η συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο και τι Εθνικέ Ελεγκτικές Αρχές επίσης πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο αυτό. Τα πρώτα βήματα έγιναν ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Eurostat προσκάλεσε τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Ελεγκτικές Αρχές για να έχουν μια ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα διαχείρισης ποιότητας. Επιπλέον, η Επιτροπή Επαφής των Εθνικών Στατιστικών Αρχών συμφώνησε να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας η οποία θα καταρτήσει κανόνες συνεργασίας ε, μεταξύ τους. Με ευθύνη για τα στατιστικά στοιχεία και για τον έλεγχο θα μπορέσω να διευκολύνω τις επαφές ε, μεταξύ των εμπλεκομένων στον τομέα αυτό, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την εξαρτησία τους. Είμαι πεπισμένος πως αυτό θα είναι επωφελές για όλους τους εμπλεκόμενους. Θα ήθελα να τελειώσω τώρα με τον προγραμματισμό. Θα λάβετε, για, την, για να το εγκρίνετε, ένα ευρωπαϊκ, σχέδιο Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος για τα έτη 2013-2017. Το πενταετές αυτό σχέδιο το οποίο συμφωνεί βεβαίως με ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, είναι μια φιλόδοξη πρόταση και θα λάβει πλήρως υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγή στατιστικών στοιχείων στην Ευρώπη. Ε, αυξημένες ανάγκες για δεδομένα, περιορισμένοι προϋπολογισμοί, ανάγκη για καλύτερη ποιότητα και μείωση του βάρους στι επιχειρήσεις και στους πολίτες. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας παρουσίασα τις βασικές προκλήσεις και προτεραιότητες για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία και κάποια νομοθετικά κείμενα τα οποία θα υποβληθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους μήνες που έρχονται. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια από καινού για να ενισχύσουμε την ε, αξιοπιστία των ε, ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων. Η δική του αξιοπιστία είναι και η δική μα αξιοπιστία. Να πω πως είμαι πεπισμένος πω η απόφαση για να συμπεριληφθούν τα στατιστικά στοιχεία στις αρμοδιότητέ μου θα ενισχύσει την ε, ανεξαρτησία τη Eurostat και θα βοηθήσει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τον Όλαφ και τις υπηρεσίε Κομισιών Αρμόδιες για τον έλεγχο. Ευχαριστώ. What I propose to do now is to continue taking προτείνω να ακούσουμε ερωτήσεις ανά τρεις, δούλεψε αυτό, διότι καμιά φορά υπάρχει αλληλεπικάλυψη. Αντί να στριμώξουμε λοιπόν την ίδια απάντηση σε ένα δίλεπτο επί τρία, έχετε περισσότερο χρόνο. Πρώτες τρεις ερωτήσεις. Φέο, Άννη Ποδηματά, Σιλβί Γκουλάχ. Και μετά θα ακούσουμε την απάντησή σας. Θα έχετε περίπου έξι λεπτά. Ο Διόγκο. Επίτροπε, ε, σε Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που ήρθατε στην Επιτροπή μας και να σας συγχαρώ και προσωπικά και εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη διέμβρηση της εντολής σας και για τις νέες ευθύνες που αναλαμβάνετε ως μέγιστος εγγυητής των ε, Ευρωπαϊκών Στατιστικών και της Eurostat. Θα ήθελα να σας κάνω μια ευθεία ερώτηση. Τον Αύγουστο του 2010 διευρύθηκαν οι αρμοδιότητες της Eurostat. Γιατί διαπιστώθηκε ότι ορισμένα στατιστικά στοιχεία για το χρέος και το έλλειμμα των κρατών ε, δεν ήταν ορθά. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος ε, στο στατιστικό σύστημα και δεν ήταν εγγυημένα πάντα τα στοιχεία. Αυτό ήταν πριν από ένα έτος και πλέον. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι έγινε και πώς θα εγγυηθείτε τώρα την αξιοπιστία ε, και την ορθότητα των στοιχείων που διαβιβάζουν σήμερα τα κράτη-μέλη, γιατί είναι εκ των όνων αυτή για να λειτουργεί το σύστημα ολόκληρο. Και θα ήθελα παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Αποδηματά, παρακαλώ. Thank you very much, uh, Sharon. Ευχαριστώ πολύ, Σάρον. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα ήθελα κι εγώ να σας συγχαρώ για τα νέα σας καθήκοντα, αλλά δεν θα σας εκπλήξει αν η ερώτησή μου αναφέρεται και συνδέεται με την πρόταση που υποβάλατε πριν από λίγες εβδομάδες για ε, τη φορολόγηση του χρηματοοικονομικού τομέα και πιο συγκεκριμένα για την εισαγωγή ενός τέλους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Uh, Έχει γίνει η πρόταση και εσείς στο ΕΚΟΦΗΝ κάνατε τις πρώτες συζητήσεις ήδη και σήμερα το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια στρατηγική θα πρέπει να καθοριστεί έτσι ώστε να ε, υπάρξει ε, αίσια έκβαση στην πρότασή σας εξετάζετε τρία διαφορετικά ενδεχόμενα. Σε επίπεδο ένωσης να εισαχθεί αυτό το τέλος ή ακόμα και σε επίπεδο κρατών μελών, αναομάδες κρατών μελών, στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας. Αλλά η πρώτη επιλογή σε πανευρωπαϊκό, πανενωσιακό επίπεδο είναι καλύτερη. Έχω να σας ρωτήσω λοιπόν τα εξής. Κατά την άποψή σας, ποια είναι η πιο κατάλληλη στρατηγική για να ενισχυθεί και να προωθηθεί αυτή η πρώτη επιλογή, η πρώτη δυνατότητα ε, να υπάρξει εισαγωγή αυτού του φόρου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεύτερη ερώτηση, εσείς προσωπικά και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανειλημμένα τονίσατε ότι ένας ε, πιο στενός ε, φορολογικός συντονισμός για αυτό το τέλος ή κάποιους άλλους φόρους ε, είναι αναπόσπαστο τμήμα ε, καλύτερου οικονομικού και δημοσιονομικού συντονισμού. Ερωτώ λοιπόν, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τι πρόκειται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι προτίθεται να κάνει για τα επόμενα μέτρα, για ε, ποια, πιο ισχυρή οικονομική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι μια ακρόαση αυτή που αφορά τις στατιστικές και όχι ε, όλο το ε, χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου. Ε, παρακαλώ να παραμείνετε ε, στο θέμα μας που έχει να κάνει με τη Eurostat και τις στατιστικές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το επόμενο ερώτημα της Σιλβί Γκουλάρ. Θα παραμείνω σε αυτό το θέμα. Πολύ καλή ερώτηση της Άννης. Ελπίζω παρόλα αυτά να απαντήσει ο Επίτροπος. Για αυτό το θέμα των στατιστικών. Ε, μπράβο, συγχαρητήρια καταρχά και χαιρόμαστε για τα μέτρα που παίρνει ο πρόεδρο Μπαρόσο και σα αναθέτει αυτέ τι αρμοδιότητες, αλλά εγώ έχω την εξή ανησυχία. Αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι ενισχύεται και είναι χρήσιμο, εντάξει, ε, ο έλεγχο, η επαλήθευση των στατιστικών, η ορθότητα, για ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα, ό,τι είναι μέσα στο σύστημα. Ενώ με το EFSF, με τα διάφορα μέτρα και ε, μηχανισμούς που εφευρίσκουμε τώρα, βγάζουμε από το ευρωπαϊκό σύστημα κάποια όργανα που είναι πλέον ιδιωτικού δικαίου και δεν τα ελέγχει ο ΔΙΣ. Και πού εντάσσονται αυτά στο θεσμικό οικοδόμημα. Εσείς πώς σκέφτεστε να επαναφέρετε λίγο την τάξη σε αυτή την αρχιτεκτονική και δεν είναι δύσκολο, δεν είναι επικίνδυνο να έχουμε διπλά στάνταρ τώρα από τη μια τον έλεγχό σας και από την άλλη όλα αυτά τα τεράστια ποσά που εκφεύγουν και της Όλαφ και της ορθότητας των στοιχείων και κάθε ελέγχου και κοινοβουλευτικού αλλά και γενικότερου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις σας. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων και ιδιαίτερα τα οικονομικά στοιχεία που δίνουν οι κυβερνήσεις. Η Eurostat έχει σήμερα εξουσίες από πέρσι συγκεκριμένα και μέχρι φέτος που είναι επαρκής για να βεβαιωθούμε ότι τα στατιστικά δεδομένα, τα στατιστικά στοιχεία που διαβιβάζονται είναι ευθύ εξ αρχής ε, σωστά. Από τα πρωτογενή στοιχεία που συλλέγονται μέχρι το τελικό στάδιο, μέχρι την υποβολή τους δηλαδή στη Eurostat, υπόκεινται σε ελέγχους, σε επαληθεύσεις από την ίδια τη Eurostat, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Είναι πραγματικό το εγχείρημα. Διπλασιάσαμε τους υπαλλήλους που ασχολούνται ειδικά με αυτά τα θέματα χωρίς να αυξηθεί γενικότερα το προσωπικό της Eurostat. Και γίνονται αυτές οι επαληθεύσεις και οι έλεγχοι σε πρώιμα στάδια. Και μεθοδολογικές επισκέψεις στα κράτη-μέλη και ελέγχονται τα στοιχεία και μάλιστα η πλήρης αλυσίδα παραγωγής στατιστικών στοιχείων. Και λαμβάνεται υπόψη αυτή η δυνατότητα που έχει και ελέγχου και επιβολής προστήμων η Eurostat όταν υπάρχουν λαθροχειρίες ε, με τα στατιστικά στοιχεία. Είναι ένα ισχυρό μέσο, ένα ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται στο μέλλον, στην πράξη και ε, στο μέλλον θα ε, ασκήσει όλο και περισσότερο και τις εξουσίες της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις προσφυγές επί παραλήψη, επί παραβιάση των ε, κανόνων που συμφωνήθηκαν. Μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο και εδώ στο Κοινοβούλιο αν δεν γίνονται αυτά σεβαστά. Αυτές λοιπόν οι νέες εξουσίες πιστεύω ότι μας δίνουν πραγματικά διασφάλιση και τα εχέγγυα ότι η ποιότητα των ε, στοιχείων που δίνουν οι κυβερνήσεις για τα οικονομικά τους είναι επαρκής. Επανέρχομαι τώρα στην άλλη μου ιδιότητα στο άλλο χαρτοφυλάκιο για τη φορολογία. Είχαμε αυτή την πρώτη συζήτηση για το φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα γνωρίζετε ότι την 9η Νοεμβρίου κάναμε και μια πρόταση για ένα ίδιο πόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και να είναι αυτό το τέλος ε, τμήμα της πρότασης αυτής και προτείνουμε να ε, μοιράζονται τα έσοδα, τα δύο τρίτα από το τέλος αυτό να πηγαίνει στο κοινοτικό προϋπολογισμό και το ένα τρίτο στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Αυτό τι σημαίνει. Είμαστε υπέρ της συμφωνίας αυτή σε επίπεδο της Ευρώπης των 27. Και στις πρώτες συζητήσεις, παρόλο που στον τύπο δημοσιεύτηκαν ε, κάποια άρθρα που λέγουν ότι τα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ διχασμένα, πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω πολύ διαφορετική ερμηνεία της πρώτης συζήτησης που είχαμε. Και οι θέσεις των κρατών μελών συγκλίνουν και για το θέμα αυτό. Και ιδιαίτερα μεταξύ των μελών της Ευρωζώνης. Βεβαίω έχουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αυτό τον καιρό, πώς να το πω, έχει τις επιφυλάξεις του για το τέλος αυτό, αλλά η συζήτηση μόλις έχει αρχίσει και οι εμπειρογνώμονές μας επισκέπτονται τις χώρες αυτές έτσι που είναι πιο διστακτικέ για την πρόταση και εξηγούν τα τεχνικά στοιχεία της πρότασης και προσβλέπω στις τεχνικές συζητήσεις στο Συμβούλιο που θα αργήσουν πάρα πολύ σύντομα την 5η Δεκεμβρίου σε ό,τι αφορά τον ε, πιο στενό συντονισμό στα φορολογικά θέματα. Με αυτό εγκρίναμε σήμερα φορολογικό συντονισμό στα πλαίσια της ετήσιας μελέτης για την, για την ε, ανάπτυξη. Γνώμη. Είναι σημαντικό το στοιχείο για τη βελτίωση και του φορολογικού συντονισμού γιατί μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να κάνουμε συστάσεις στα κράτη-μέλη. Τι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν, ε, έτσι φορολογικές, Έχουμε μελετήσει και υπολογίσει τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών και είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις. Εδώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό μέσο ε, που θα οδηγήσει σε πιο στενό ε, συντονισμό των φορολογικών πολιτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λογοδοσία των ευρωπαϊκών μηχανισμών. Τώρα, έχουμε ένα μηχανισμό σήμερα που λειτουργεί και συνδέεται στο, τμήμα του που αφορά τον κοινοτικό προπολογισμό ε, υποβάλλεται σε ελέγχους οικονομικούς από το ελεγκτικό συνέδριο. Και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ESM, προβλέπει την ανάγκη μάλιστα εξωτερικών οικονομικών ελέγχων αυτού του μηχανισμού. Βεβαίως τώρα γίνεται και μια συζήτηση για το ποιος θα πρέπει να κάνει αυτούς τους οικονομικούς ελέγχους. να είναι κάποιος εξωτερικός ιδιώτης ή δημόσια αρχή. Δεν έχει λήξει αυτή η συζήτηση, δεν έχει καταλήξει, αλλά είναι σαφές ότι οι συνάδελφοί μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι βεβαίως υπέρ της πλήρους λογοδοσίας και διαφάνειας και σε αυτούς τους μηχανισμούς. Ε, thank you very much. Um, ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνω με τις επόμενες ερωτήσεις η Σουίνμπερν, Φιλίπ Λαμπέρτς, που θα συνδυάσει τις δύο ερωτήσεις του, νομίζω, και εσείς και αν θέλετε, και μετά ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, με ενδιαφέρον άκουσα για τα νέα σας καθήκοντα και την ανεξαρτησία της Eurostat και πραγματικά ελπίζω να μπορέσετε να επιτύχετε τους στόχους ε, τους οποίους αναφέρατε σήμερα καιρός νομίζω ήταν να έχουμε λίγη περισσότερη εμπιστοσύνη στη λειτουργία της ε, Eurostat και αυτό το οποίο μας είχε πει πριν από ένα χρόνο η Eurostat ήταν πως ε, υπάρχει πλέον απέτηση για οποιοδήποτε μέσο χρηματοδότησης εκτός ισολογισμού να δηλώνεται από τα κράτη-μέλη στη Eurostat και συγκεκριμένα με ενδιαφέρει το πως οι δεσμεύσεις του EFSF, ε, δηλαδή το μεγαλύτερο τέτοιο όχημα ειδικού σκοπού θα εμφανιστεί στους ε, ισολογισμούς των κρατών μελών. Φαντάζομαι θα έχετε λίγο χρόνο να το σκεφτείτε. Και το δεύτερο ερώτημά μου ε, δεν ε, θα το ανέφερα, αλλά μια που το θίξατε νομίζω λογικό είναι. Θα ήθελα εγώ να αφιερώνετε τόσο περισσότερο χρόνο μπορείτε στο νέο σας ρόλο και να μην χρειάζεται να ασχολείστε πλέον με τον Ευρωπαϊκό Φόρο ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και οπωσδήποτε δεν είχα αμφιβολία πω ο Υπουργό Οικονομικών μα θα έλεγε όχι και πάλι όχι και μετά όχι. Και δεδομένου του ότι τρία κράτη-μέλη έχουν πει όχι, δηλαδή Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και Τσεχία, ανησυχώ λίγο για το ότι θα αφιερώνεται χρόνο σε κάτι τέτοιο όταν απαιτείται ομοφωνία. Ε, μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε πως θα αφιερώνετε περισσότερο χρόνο στη γύρω στα στο μέλλον. Ναι. Φιλίπ. Ναι, κύριε Επίτροπε, θέλω <coughs> πρώτα χαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε για το EGS, το αναφέρετε. Νομίζω ότι φτάνει το τέρμα και το βλέπουμε για τη στα λοιπόν. είδα την απάντησή σας στο, στα γραπτά ερωτήματα όσον αφορά τους δείχτες τους ποιοτικού των εισοδημάτων βασίζεται στον αριθμό ανθρώπων που κινδυνεύουν τη φτώχεια. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ε, όλης υποθέσεως. Θα έπρεπε να έχουμε καλύτερη ένδειξη της σταδιακής διανομής του ε, κατανομής του εισοδήματος. Δεν είναι ότι μας ενδιαφέρουν μόνο οι φτωχοί, αλλά και οι υπερβολικά πλούσιοι. Ε, πρέπει να βρούμε πού βρισκόμαστε και πώς ε, αποδίδουμε ξέροντας ότι τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι ε, πιο ισότιμες κοινωνίες αποδίδουν καλύτερα. Δηλαδή μιλάμε πιο ισότιμες όσον αφορά το εισόδημα. Δεύτερον, κάτι που δεν καλύφθηκε από την, προφορή, από την γραπτή ερώτηση, η ανεργία. Ε, ίσως θα με ενημερώσετε γιατί ίσως δεν γνωρίζω τόσο καλά τα στατιστικά, τα παρόντα στοιχεία της Eurostat. Η Eurostat πώς μπορεί να αξιολογήσει το υποκείμενο επίπεδο, όχι μόνο τη ανεργία, αλλά τη υποαπασχόληση επίση. Ξέρουμε καμιά φορά ίσω να φαινόμαστε αρκετά καλά όσον αφορά την απασχόληση, αυτό δεν ισχύει σήμερα, αλλά να υποφέρουμε πολύ ε, λόγω μη επιλεγμένη μερική απασχόληση κλπ. Σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, πού βρισκόμαστε, υπάρχουν εφήμε σύμφωνα με τι οποίε η πραγματική ανεργία ε, είναι κοντά στο 20% αν τα υπολογίσουμε αυτά και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σα. Και συνεχίζει εκτό μικροφώνου πλέον ο ο κύριος Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση, κύριε Σεμέτα, με βάση τα καινούργια σας καθήκοντα. Σας εύχομαι ειλικρινά να τα καταφέρετε. Η ερώτησή μου έχει να κάνει μέχρι πού φτάνει η δική σας ευθύνη σχετικά με τη Eurostat. Αναφέρομαι στον όρο Greek Statistics που από ό,τι φαίνεται όμως ήταν μια συνηθισμένη πρακτική από πολλές χώρες να αλλοιώνουν στοιχεία για το ΑΕΠ και η Eurostat να το ανέχεται. Αναζητούνται σε μια τέτοια περίπτωση, δεν σας εύχομαι να σας συμβεί, αναζητούνται και προσωπικές ευθύνες στον Επίτροπο που εποπτεύει τις Eurostat σε τέτοια περίπτωση και τι σημαίνει αυτό. Και η δεύτερη ερώτηση, απλή για την ιδιότητά σας που εξακολουθείτε να έχετε, φορολογικού περιεχομένου. Η ελληνική κυβέρνηση έβαλε φόρο στα ακίνητα ανάγκασε την υπηρεσία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας να εισπράττει αυτό τον κρατικό φόρο. Με απειλή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Η ερώτηση. Είναι συμβατή με τέτοια πρακτική με την κοινοτική νομοθεσία. Δηλαδή πάροχος υπηρεσιών να εισπράττει κρατικούς φόρους. Ευχαριστώ θα κάνει ό,τι μπορεί ο κύριος Επίτροπος με τι ερωτήσει. Ήρθε προετοιμασμένος για στατιστικά στοιχεία και όχι για ερωτήσεις ε, φορολόγηση. Ε, έχετε το λόγο. Ε, για όσον αφορά τη φορολόγηση, μπορώ να μιλήσω και χωρίς πολλή προετοιμασία. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε το EFSF. Και σε σχέση με τα στατιστικά. Η χρηματοδότηση του FSF ξαναδρομολογείται προς το δημόσιο χρέος του κράτη και υπολογίζεται ως τέτοιο. Όλες οι πληροφορίες που δίδονται το δημόσιο χρέος αποκαλύπτονται και για το FSF. Άρα υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το δεύτερο ερώτημα σας. Θα σας απογοητεύσω αλλά θα εξακολουθώ να, μιλήσω για, να μιλάω για το φόρο για τις χρηματοσυντικές συναλλαγές και να τον υποστηρίζω ένθερμα και ελπίζω να έχω επαρκή χρόνο για όλα τα μέρη του χαρτοφυλακίου μου και δεν θα υποφέρουν τα στατιστικά στοιχεία λόγω της εργασίας μου για, τον, για τη φορολόγηση χρηματοσυντικών συναλλαγών. Μετά το θέμα για το θέμα αυτό της ηλεκτρικής ενέργειας Καταλαβαίνω αυτά που μου είπατε για τη διακοπή του ηλεκτρικού. Και τα στοιχεία για την ηλεκτρική ενέργεια και τους δείκτες Υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων. Έχουμε Συμβουλευτική Επιτροπή για τα Ευρωπαϊκά Στατιστικά Στοιχεία, όπου οι χρήστες των στατιστικών στοιχείων και η παραγωγή στατιστικών στοιχείων και οι στατιστικολόγοι οι ίδιοι συναντώνται και αναλύουν και τις νέες ανάγκες, τις ανάγκες των νέων χρηστών και τα θέματα που άπτονται με την παραγωγή στοιχείων. Και τα νέα στατιστικά στοιχεία φέρουν και βάρος στους χρήστες. Θα τα συζητήσουμε και αν υπάρχει ανάγκη βελτίωσης αυτού του τομέα των στατιστικών στοιχείων μπορεί να συζητηθεί το θέμα για την απασχόληση. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, επικαιροποίησε το σύστημά της η Ευρωστάτ των δικτών για την ανεργία. Συμπεριλήφθησαν τρεις νέοι δείκτες στο σύστημα και ένας δίκτης για την υποαπασχόληση συμπεριελήφθη. Στους χρήστες θα δοθούν οι πληροφορίες μέσω της εκτεταμένης αυτής βάσης δεδομένων της Eurostat και όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου καλούνται να χρησιμοποιήσουν στο βαθμό του δυνατού όσο θέλουν τη βάση δεδομένων. Το ερώτημα μετά για τις ευθύνες που έχω απέναντι στην Eurostat, να τονίσω ότι χρειαζόμαστε ανεξάρτητο, ανεξάρτητη στατιστική υπηρεσία που λαμβάνει τις αποφάσεις της βάσει επαγγελματικής ανεξαρτησίας, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των αποφάσεών της. Στο χαρτοφυλάκιά μου έχω την Όλαφ, η οποία έχει παρόμοιο καθεστώς, είναι ανεξάρτητη υπηρεσία, ανεξάρτητος φορέας, Υπάρχει, έχω υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου υπό τις ευθύνες μου και εκεί και αυτή η δομή είναι ανεξάρτητη Ξέρω συνεπώς πώς να χειρίζομαι ανεξάρτητους φορείς. Δεν είναι εύκολο το έργο. Νομίζω ότι συνδυάζοντας την εμπειρία από άλλα τμήματα του χαρτοφυλακίου, από άλλους τομείς, το αποτέλεσμα το τελικό θα είναι καλό και για το συγκεκριμένο θέμα. Το ερώτημα για τη φορολόγηση όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού πρέπει να σας πω ότι οι φορολογικές αρχές στην Ελλάδα, η φορολογήση στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι, η αντιμετώπιση φορολογής στην Ελλάδα είναι σοβαρό πρόβλημα και εξακολουθεί να είναι και η task force που δημιουργήσαμε για να βοηθήσει και να παράσχει τεχνική αρρωγή στην Ελλάδα ασχολίζεται και με την εφορία, με θέματα φόρων από τις ελληνικές αρχές εξαρτάται η σύσταση, η δημιουργία του συστήματος αυτού που συλλέγει με τον καλύτερο τρόπο τον φόρο, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη το πόσο μεγάλα ελλείμματα υπάρχουν στην Ελλάδα και πόσο χρειάζεται η βελτίωση της ίσπραξης φορολογικών εσόδων. Αν η μέθοδος που εισήχθη στην Ελλάδα επιτρέπει τη συλλογή φόρων αποδοτικότερα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, τότε είναι ευπρόσδεκτη αυτή η προσέγγιση. Δεν μπορεί παρά να είναι ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ πολύ. Δύο μόνο συναδέλφους έχω που θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Αν θέλει κι άλλος να ρωτήσει, η Μάριαν. Αρλίν, λοιπόν. Σάντελ ο Καντράουι και μετά η Μαριάν. Ε, um, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να μιλήσω για τα στατιστικά στοιχεία. Θέλω να μάθω τι στοιχεία συλλέγεται για φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, γιατί δεν έχω βρει ε, στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν παγκόσμια και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έλλειψη των στοιχείων σημαίνει πως χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για αυτό το ζήτημα, το οποίο βεβαίως κοστίζει έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μυστικότητα κάποιων διμερών συμφωνιών... Ε, σημαίνει πως είναι δυσκολότερο να βρεθούν τα στοιχεία. Οπότε, τι προσπάθειες θα καταβάλλετε για να έχουμε περισσότερη διαφάνεια, για να έχουμε μια ιδέα για την κλίμακα, την τάξη του προβλήματος. Και να σας ρωτήσω, η Eurostat θα κοιτάξει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο για τις χώρες οι οποίες ε, μπορεί να επιλέξουν να εισαγάγουν ένα τέτοιο φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, είτε είναι η Ευρωζώνη είτε κάποιε άλλε. και να μάθω τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στο City του Λονδίνου, αν μείνει εκτός ενός τέτοιου φόρου. Σαΐντ, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, συνάδελφε, θέλω να αναφερθώ στο τελευταίο ερώτημα της Αρλίν. Νομίζω πως είναι ουσιαστικό Είμαστε σε μια κατάσταση όπου φαίνεται πως κάποια κράτη-μέλη η συλλογή των φόρων ε, λαμβάνει χώρα πάρα πολύ άσχημα. Πρέπει να συλλέξουμε υλικό και να το ερμηνεύσουμε επίσης και το ερώτημά μου είναι βλέπετε οι αρμοδιότητες ε, οι οποίες θα λάβετε να έχουν κάποιες δυνατότητες να υπάρξει κάποια συγκριτική αξιολόγηση, να οδηγήσετε σε κάποια καλύτερη εξέλιξη αυτών των πραγμάτων. Και βεβαίως, επειδή είστε και υπεύθυνο για την φορολογία, όσον αφορά κάποια... Πώς το βλέπετε να λάβετε κάποια πρωτοβουλία όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων για φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή για να γίνει αυτή δυσκολότερη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπω πως ο κύριος Κιούτας έφτασε. Θα ακούσουμε και αυτόν άρα. Μαριάν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, διάβασα διάφορες ιστορίες ε, στον ε, τύπο για στατιστικά στοιχεία και την ποιότητά τους που λένε πως εάν δει κανείς ε, σειρές στατιστικών στοιχείων για ελλείμματα προϋπολογισμού και, ε, και χρέους πως υπάρχουν εκεί πέρα πάρα πολλές μεγάλες αποκλήσεις ε, και αυτό θα πρέπει να αποτελήσει αντικείμενο ερώτηση. Εγώ δεν ξέρω τίποτα περί στατιστικής, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε από τα πανεπιστήμια, εμφανίζονται αυτά στον τύπο και είναι ζητήματα τα οποία επανεμφανίζονται. Το ερώτημά μου λοιπόν προς σας είναι τα γνωρίζετε αυτά, ε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά ή είναι απλά μπουρδες. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο παρακαλώ να μας το πείτε, ε, να τα ακούσουμε από το δικό σας στόμα. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, γνωρίζω βεβαίως πως η συζήτησή μας αφορά τα στατιστικά στοιχεία, αλλά μια που είναι εδώ πέρα ο κύριος Επίτροπος, θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η απόψή του για τη φορολογική εναρμόνιση στα κράτη-μέλη. Θεωρώ πως ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες διμερείς συνεννοήσεις όπως η γαλλογερμανική ας πούμε που είναι κάπως περιορισμένες. Οπότε πιστεύω πως μια κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις θα μπορούσε να υιοθετηθεί αλλά η συμμετοχή σε αυτή θα έπρεπε να είναι προαιρετική και για τα κράτη-μέλη και για επιχειρήσεις και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια βήματα προβλέπετε να γίνουν εάν θέλετε να συνεχίσουμε με την εναρμόνιση της ε, άμεσης φορολογίας στα κρατημέλη που εγώ πιστεύω πως είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Νομίζω πως τελείωσαν οι ερωτήσεις. Προφανώς ε, ναι. μας ενδιαφέρει πιο πολύ η φορολογία παρά τα στατιστικά στοιχεία. Δυστυχώς η φορολογία εξακολουθεί να είναι πιο ενδιαφέρουσα από τα στατιστικά στοιχεία, αλλά ελπίζω τα επόμενα χρόνια να αφιερώσουμε ίσο χρόνο στα δύο στην Επιτροπή αυτή. Τώρα όσον αφορά τη στατιστικά στοιχεία, πρώτα απ' όλα για τη συνεργασία μεταξύ Ταξούντ και Eurostat. Από κοινού παράγουν ένα έγγραφο στο οποίο αξιολογούν τα στατιστικά στοιχεία για την φορολογία στα κρατημέλη είναι ένα μεγάλο έγγραφο όπου μπορείτε να δείτε τι γίνεται στα συστήματα τα φορολογικά των κρατών μελών. Αλλά δυστυχώς στατιστικά στοιχεία για φοροαποφυγή δεν είναι διαθέσιμα. Δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογή στοιχείων μπορούμε να το υπολογίσουμε κάπως εμέσως γιατί τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των εθνικών λογαριασμών πρέπει να κάνουν έναν υπολογισμό της λεγόμενης ε, παραοικονομίας. Οπότε από αυτά μπορούμε να εκτιμήσουμε εμέσως ποια θα ήταν τα αποτελέσματα συλλογή των φόρων, αλλά δεν συλλέγονται τέτοια στατιστικά στοιχεία, αλλά είναι ενδιαφέρον ε, θέμα, το οποίο οπωσδήποτε θα συζητήσω με τους ειδικούς στη Γυροστάτ, γιατί όπως εξημάνατε η φοροαποφυγή είναι πολύ σημαντικό θέμα και εάν ε, μπορούμε να συλλέξουμε φόρους καλύτερα από ό,τι το κάνουμε τώρα, δεν θα έχουμε ανάγκη να αυξήσουμε το επίπεδο των φόρων. Οπότε το θέμα αυτό είναι κορυφαία προτεραιότητα για το πρόγραμμα του επομένου έτους ε, της φορολογίας, να δούμε φορολογικούς παραδείσους, ε, την ε, μη φορολόγηση κτλ. και θα συνεργαστώ με την Επιτροπή σας. Όσον αφορά στατιστικά στοιχεία, όσον αφορά στατιστικά για τον φόρο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και την πιθανή εισαγωγή του. Σε πιθανή εισαγωγή του σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, βεβαίως δεν ε, υπάρχει ακόμα αυτός ο φόρος, οπότε δεν μπορούμε να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία. η αξιολόγηση αντικτύπου ε, είχε γίνει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν μπορώ να σας πω... Ε, είναι αδύνατο να σας πω αυτή τη στιγμή ε, στατιστικά δεδομένα γιατί δεν υπάρχει ο φόρος. Μετά, όσον αφορά τα ζητήματα της ε, φοροαποφυγής και της ανταλλαγής πληροφοριών. Ξέρετε πως έχουμε το σύστημα το Eurofisk για την ανταλλαγή πληροφοριών για ζητήματα ΦΠΑ και ο ΦΠΑ είναι ένας τομέας όπου η απάτη είναι σημαντικό πρόβλημα. Το Δεκέμβριο θα υποβάλουμε μια στρατηγική για το μελλοντικό ΦΠΑ όπου το στοιχείο καταπολέμησης απάτης θα είναι πολύ έντονο και βεβαίως εξετάζουμε και τις δυνατότητες ε, βελτίωσης. Βεβαίως το σύστημα γυροφίσκ μόλις δημιουργήθηκε οπότε πρέπει να επιταχύνουμε την ανάπτυξή του για να επωφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα αυτού του νέου συστήματος, αλλά βεβαίω αναμένω τις βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα, γιατί το Eurofisk μας επιτρέπει το να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ κρατών μελών και στον τομέα της ε, απάτης ε, της φορολογικής του ΦΠΑ η, η ταχύτητα ανταλλαγής πληροφοριών έχει μεγάλη σημασία οπότε όταν θα λειτουργεί το Eurofisk πλήρως νομίζω πως η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί σημαντικά κατόπιν, αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση ε, μιλήσετε για αναθεώρηση στατιστικών σειρών. Ε, κοιτάξτε, είναι σύνηθες να γίνεται αναθεώρηση των στατιστικών σειρών. Είναι μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται στη στατιστική όταν ε, έχουμε νέες εξελίξεις σε κάποιον τομέα της στατιστικής και για να διατηρηθεί η συγκρισιμότητα των στατιστικών σειρών υπάρχει ανάγκη αναθεώρησής τους. Βεβαίως υπάρχουν ε, και αναθεωρήσεις ε, π.χ. έχουμε παρουσιάσει στην Άνοιξη και το Φθινόπωρο. Ε, και το Φθινόπωρο έχουμε ακριβέστερα στοιχεία ε, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να συλλέξουμε ε, πλήρεις πληροφορίες και βεβαίως ε, η αναθεώρηση αυτή μεταξύ άνοιξης και φθινοπόρου είναι και ένα στοιχείο ποιότητας ακριβώς για να έχουμε αυτή την αλλαγή, η οποία βεβαίω θα πρέπει να είναι όσο δυνατόν μικρότερη από την άνοιξη ε, στο φθινόπωρο, αλλά κάποιε αλλαγέ είναι αναπόφευκτες λόγω της διόρθωση των στατιστικών δεδομένων. Και το τελευταίο ερώτημα για την φορολογική εναρμόνιση και την κοινή φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις. Μπορώ να πω πως Έχουμε ένα σύστημα έμεσων φόρων, ΦΠΑ, φόροι κατανάλωσης, όπου υπάρχει πολύ περισσότερη, ε, πολύ μεγαλύτερη εναρμόνιση και απαιτείται πολύ μεγαλύτερη εναρμόνιση και τυποποίηση. Και αυτό θα το δούμε στην επόμενη ανακοίνωση για το μέλλον του ΦΠΑ γιατί η τυποποίηση εάν γίνει πολύ καλύτερη, θα μειωθεί και το διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις. Και θα αντιμετωπίσουμε την απάτη του ΦΠΑ, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τους άμεσους φόρους, η κοινή φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις είναι πρόταση της εσωτερικής αγοράς εάν ε, μπορέσουμε να συμφωνήσουμε από αυτού και ε, εγώ βλέπω κάποιες ε, σοβαρές εξελίξεις στον τομέα αυτών τώρα που τα κράτη-μέλη συζητάνε την ίδια την φορολογική βάση γιατί είναι προαπαιτούμενο να συμφωνήσουμε με τις φορολογικές βάσεις για να μπορέσουμε αργότερα να συμφωνήσουμε σε μια ενοποίηση και μια επίσημη κατανομή που είναι πιο ε, ουσιαστικά ζητήματα. Τώρα, γιατί προτείνουμε κάτι το προαιρετικό, γιατί υπάρχει ποικιλομορφία στα κράτη-μέλη και αυτό το προτείνουμε σε ένα 28ο καθεστώς, εάν θέλετε. Ε, υπάρχει και σε άλλους τομείς και λαμβάνουμε υπόψη το ότι υπάρχουν μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, ε, επιχειρήσεις οι οποίες ε, δραστηριοποιούνται σε κάποιες μικρούς, μικρές περιοχές και δεν έχει νόημα να δραστηριοποιηθούν διασυνοριακά. Οπότε αν θέλουν να μείνουν ε, στο εθνικό σύστημα, νομίζουμε πως αυτό είναι θεμητό. Το ερώτημά σας αφορούσε τον συντονισμό μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Δεν βλέπω εγώ κανένα πρόβλημα με το να θέλουν κάποια κράτη-μέλη να πάνε παραπέρα με βάση την ε, πρόταση αυτή για κοινή φορολογική βάση. Αν συμφωνήσουμε σε επίπεδο Ένωση και μετά κάποια κράτη-μέλη θέλουν να εναρμονίσουν τα συστήματά τους, ε, λαμβάνοντας υπόψη πως η Γαλλία και η Γερμανία είναι μέλη της Ευρωζώνης, τα μεγαλύτερα μέλη της Ευρωζώνης, ε, δεν βλέπω εγώ κανένα πρόβλημα. θα μπορούσε δε να αποτελέσει η κοινή αυτή φορολογική βάση, τέλεια βάση για κάτι τέτοιο. Τελείωσαν οι ερωτήσεις. Να σας πω λοιπόν ότι η έκθεση για το, ίσα, για το 2020 θα δημοσιευθεί σύντομα. Έχει αποσταλεί στη γραμματεία όπου κάνω κάποια μυστήρια πράγματα πριν δημοσιευθεί. Θα το δείτε το κείμενο σύντομα. Και θέλω εκεί να ελαχιστοποιήσω τις ε, εξαιρέσεις και παρεκκλήσεις, να δούμε πώς θα πάει μαζί με κάποια άλλα πράγματα. Και όπως ίσως ε, ήδη γνωρίσετε, ε, κλέψαμε κάπως ε, κάποια που υπόθηκαν εξαρτησία των στατιστικολόγων και το βάλαμε στη δέσμη των 6 μέτρων, ε, στο six pack και θα το υποστηρίξει αυτό η Επιτροπή. Όταν θα συζητηθεί ανακοίνωση που αναμένουμε από εσά. Προσβλέπουμε συνεργασία μαζί σας για τα στατιστικά στοιχεία, τα κακά μαντάτα είναι ότι πιθανότατα αυτό σημαίνει ότι ε, θα είμαι εγώ ε, που θα σας περιμένει. Ευχαριστώ που ήρθατε, ευχαριστώ που απαντήσατε και τις ερωτήσεις για τους φόρους. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει και ο Επίτροπος. Εργάστηκα για τα στατιστικά στοιχεία. Επί 7 χρόνια εργάστηκα σε στατιστική υπηρεσία, ήμουν επικεφαλής και ξέρω πόσο σημαντική είναι η ανεξαρτησία των στατιστικών φορέων. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να εξασφαλίσω την ανεξαρτησία τη Ευρωστάτ όχι μόνο σε Ευρωστάτ αλλά και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών και πιστεύω ότι αυτό θα εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα των επισήμων στατιστικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, λέει ευχαριστώ όλους. Έληξη συνεδρίαση, καλό σας βράδυ.